Dear colleague, please sit down. We have to... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα και έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Ενεργέτικοι senza uno stretto collegamento con le evoluzioni Καλημέρα σας. Έχουμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο και ο κόσμος της ενέργειας ε, περνά βαθιές αλλαγές. Ε, είναι οι συνέπειες αυτού του σενάριου που είναι υπό εξέλιξη και είναι όλα αυτά ε, αισθητά στην καθημερινή μας ζωή και στις οικονομίες των χωρών μας. Πρόσφατα είδαμε στην Ιαπωνία το πυρηνικό ατύχημα που όθησαν ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όπως η Γερμανία και η δική μου χώρα να ξανασκεφτούν, να αναθεωρήσουν τις ενεργειακές τους πολιτικές και αυτό μας οδηγεί σε αναθεώρηση και εξέταση όλων αυτών των υποθέσεων. Το μελλοντικό μείγμα ενεργειακού ανεφοδιασμού τίνει να τροποποιηθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον με βάση αυτά τα δεδομένα. Και υπάρχουν διάφοροι που πιστεύουν ότι η συμβολή του φυσικού αερίου μεταξύ των άλλων ενεργειακών πηγών μπορεί να επαναξιολογηθεί. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να είναι υποεξέλιξη και διαδικασίες εκδημοκρατισμού που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές ε, του 2001, λέει ο μιλητής, και βρίσκονται σε ε, εξέλιξη ακόμα στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Αυτά όλα μας οδηγούν ακόμα μια φορά να σκεφτούμε πιο σοβαρά την ασφάλεια του ε, ανεφοδιασμού σε ενέργεια και μας υποχρεώνουν να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ανεφοδιασμού μας. Γι' αυτό και μαζί με τον συνάδελφο Ρελ, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ήτρε, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση από κοινού με τις ε, δύο επιτροπές μας που έχουν εργαστεί τα τελευταία χρόνια πολύ εντατικά για αυτά τα θέματα αλλά είναι απαραίτητο αυτή η εργασία να αναπτυχθεί και να συνεχιστεί λαμβάνοντας υπόψη και τους εμπορικούς δεσμούς που έχουν οι χώρες μας με τις χώρες προμηθευτές ενέργειας στην Μεσογειακή Λεκάνη. Η ΕΝΗ είναι η έκτη παγκόσμια πετρελαϊκή εταιρεία. Είναι η πρώτη για την πώληση του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ο πρώτος, η πρώτη στην Αφρική. Από την δεκαετία του 50 έχει εμπορικές συναλλαγές με τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής όπως η Λιβύη, την Ισία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Εμέν, το Κατάρι, το Ιράν, το Ιράκ και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Σκαρόνη θα μας παρουσιάσει τα θέματα και έχει δώσει και ένα τίτλο στην παρέμβασή του. Εγώ θα ήθελα ωστόσο να προτείνω ένα προβληματισμό και για τη συζήτηση που θα γίνει στη συνέχεια και θα ήθελα να γνωρίζω την μαρτυρία του πώς μια τόσο μεγάλη και σημαντική εταιρεία που έχει αυτό τον ηγετικό ρόλο για τον ανεφοδιασμό στην Βόρεια Αφρική, πώς διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση που είναι τόσο περίπλοκη. και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής, καθώς και η δική μας συμβολή, ώστε να έχει αίσια έκβαση το θέμα του ανεφοδιασμού για τις χώρες μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Ορέλ για να κάνει και εκείνο την εισήγησή του. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σκαρόνη, καλώς ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτη ε, παρατήρηση που έχει, αφορά τη διερμηνία. Η γερμανική διερμηνία δεν λειτουργεί καλά. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, λέει ο μιλητής. Ίσως μπορεί κάποιος να το ελέγξει, παρακαλώ, και να το ρυθμίσει. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους θερμά εδώ. Ο συνάδελφος Αλπεπτίνη ήδη ανέφερε ότι αποφασίσαμε ε, να μην ε, συζητάει κάθε επιτροπή ξεχωριστά το θέμα αυτό, αλλά ε, μαζί οι δυο μας επιτροπές να συζητήσουν το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα ενεργειακής πολιτικής μεγάλης σημασίας, είναι όμως και θέμα εξωτερικής πολιτικής μεγάλης σημασίας και γι' αυτό μάλλον είναι σοφό να μην εργάζεται ο καθένας ξεχωριστά, αλλά να συνεργαστούμε ώστε οι δύο επιτροπές μας μαζί να καλέσουν κάποιους σημαντικούς εμπειρογνώμονες. Και σήμερα καταφέραμε πράγματι να καλέσουμε πολύ σημαντικούς εμπειρογνώμονες. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σκαρόνη που είναι διευθυντής στην ΕΝΗ που είναι σημαντική παρουσία στο ενεργειακό πεδίο και γι' αυτό είναι και σημαντικός συνομιλητής για μας. Το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ότι και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και σε επίπεδο ενεργειακής πολιτικής ε, σημαντικό είναι να μην κάνει κανείς τίποτα βιαστικά αλλά να ακούσει προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες και κατόπιν να λάβει κανείς αποφάσεις. Η Επιτροπή μα είναι υπεύθυνη για την η Επιτροπή μου είναι υπεύθυνη για την ενέργεια και μπορώ να σα πω ότι πολύ συχνά κινδυνεύουμε να πάρουμε βιαστικέ αποφάσει χωρί να ακούσουμε τι απόψει των διαφόρων μερών. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα, που είναι εδώ οι συνάδελφοι. Ε, κρίμα που δεν μπόρεσαν όλοι οι συνάδελφοι να είναι παρόντες ώστε να ακούσουν ε, πληροφορίες, τις πληροφορίες αυτές. Ε, αυτά αρκούν για εισαγωγή. Θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε τις εμπειρογνώμονες και γι' αυτό δίνω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Παόλο Σκαρόνη. Καλώς ήρθατε θερμά εδώ στο Κοινοβούλιο. Και σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε μαζί μας και να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Buongiorno a Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρη για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ε, σημερινή ακρόαση. Μια ανακρόαση που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, δεδομένη σε αυτή τη φάση αλλαγών και μεγάλη αβεβαιότητα που διανύουμε. Θα ήθελα να σα μιλήσω για το πώ η ΕΝΗ, η δική μου διαχειρίζεται την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Είμαστε η πρώτη παραγωγή στην Αίγυπτο, στην Λιβύη, στην Αλγερία και στην Τινησία. Η θέση μας λοιπόν στη Βόρεια Αφρική είναι πολύ σημαντική και έπειτα να σας ε, πω ποια είναι η δική μας ερμηνεία για τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης και τι κάνουμε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια της ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο για την Ευρώπη. Στη Βόρεια Αφρική υπάρχουν ε, διάφορες καταστάσεις πυδινητικής ή καθημερινής ε, αστάθειας που εξελίσσονται επίσης καθημερινά και χρειάζεται να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι χώρες αυτής της περιοχής παίζουν σημαντικό ρόλο για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη που βρέχονται από τη Μεσόγειο και που εξαρτώνται από το βορειοαφρικανικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό τα όσα συμβαίνουν στην Αλγερία και στην Αίγυπτο που παράγουν το 90% του βορειοαφρικανικού φυσικού αερίου έχει άμεσες επιπτώσεις στο ενεργειακό, ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Και επίση αυτά που συμβαίνουν ε, στην Τινησία είναι πολύ σημαντικά γιατί μέσα από την ε, τινησιακή επικράτεια περνά ο αγωγός TTPC που επιτρέπει στο αλγερινό φυσικό αέριο να φτάσει στην Ιταλία, όπου αποτελεί πάνω από το 1 τρίτο του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Μετά από την αναχώρηση του την Προέδρου Μπεναλή στις 14 Ιανουαρίου, διαπιστώσαμε μείωση της ροής του φυσικού αερίου κατά 40%. Αλλά ευτυχώς η κατάσταση επανήλθε στο κανονικό μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο ήταν μια πολύ ανησυχητική εικόνα για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση η αστάθεια στην νησία όσον αφορά την παροχή του ελγερινού φυσικού αερίου. Στην Αίγυπτο δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το κανάλι του Σουέζ μέσω του οποίου περνά 10% του υγρού φυσικού αερίου του κόσμου. Όμως η κατάσταση δεν έχει ακόμα ηρεμήσει. Στις 5 Φεβρουαρίου μια έκρηξη στον σταθμό συμπίωσης του ΕΛΑΡΗΣ στο Σινά αυτή η, αυτός ο σταθμός συμπίκνωσης είναι το κέντρο ας πούμε, της συγκέντρωσης του Αιγυπτιακού φυσικού αερίου ε, δημιούργησε προβλήματα για την Ιορδανία και τη Συρία ε, χρειάστηκαν πέντε εβδομάδες για να διορθωθούν οι ζημιές και μετά από πέντε εβδομάδες υπήρξε άλλη μια έκρηξη και μετά από τις βόμβες υπάρχει και δικαστικό θέμα γιατί υπάρχει αντιπαράθεση ενώπιον των Αιγυπτιακών ε, δικαστηρίων και αυτό είναι ε, μία από τις καταγγελίες, μία από τις κατηγορίες κατά του Μουμπάρακα και της οικογένειάς του ότι το αιγυπτιακό φυσικό αέριο πολέθηκε σε πολύ χαμηλές τιμές στο Ισραήλ. Για την Τινησία και την Αλγερία ξεκίνησε μια διαδικασία χωρίς μεγάλα προβλήματα προ τον εκδημοκρατισμό. Η κατάσταση αυτής της χώρας με ανησυχεί πολύ λιγότερο σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν φυσικά του τελευταίους τέσσερι μήνες στην ε, Λιβύη και στις μη αισιόδοξε προβλέψεις όσον αφορά την εξέλιξη της στρατιωτικής και πολιτικής κατάστασης τη χώρα αυτή. Η Λιβύη παρέχει το 1 τέταρτο των εισαγωγών ακατέργαστου πετρελαίου για την Ιταλία. Είναι ο πρώτος μας προμηθευτής. Για την ανεφοδιασμό σε πετρέλαιο δεν έχουμε πρόβλημα για να σας πω την αλήθεια. Μπορούμε να το πάρουμε και σε ποσότητα και σε ποιότητα να το αντικαταστήσουμε από άλλους προμηθευτές και θα πρέπει να σας πω ότι ο ΠΕΚ έπαιξε ηγετικό ρόλο και μπόρεσε να αντικαταστήσει κυρίως την ποιότητα του ακατέργαστου πετρελαίου για να μην μείνουν τα δηληστήρια χωρίς τα προϊόντα τα οποία συνήθως επεξεργάζονται. Πολύ πιο λεπτή βέβαια είναι η κατάσταση όσον αφορά το φυσικό αέριο το Φεβρουάριο χρειάστηκε να διακόψουμε την παροχή μέσω του αγωγού Green Stream που συνδέει τη Λιβύη με τη Σικελία. Μιλάμε για 10 δις κυβικά μέτρα αερίου. Δηλαδή το 30% των αναγκών της Ιταλίας, γιατί η Ιταλία είναι μέγας καταναλωτής αερίου καταναλώνει τόσο όσο και η Αγγλία, δηλαδή 90 δις τετραγωνικά, ε, κυβικά μέτρα το χρόνο. Αυτή την έλλειψη του λιβικού αερίου την, αντι, ε, αντισταθμίζουμε με άλλες υποδομές και το φυσικό αέριο που μας δίνεται από άλλες, άλλου τύπου συμβάσεις, take or pay. Και έτσι ε, κάνουμε ανάλογα με τις ανάγκες ε, της στιγμής. Χάρη στις ε, πολιτικές που ασκήσαμε τα περασμένα χρόνια έχουμε διαφοροποιημένες παροχές, το βλέπετε στα slides, στις διαφάνειες, και είναι δύο χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια εισάγαμε πάνω από το ίμιση του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούμε στη χώρα μας. Ε, Αλγερινό φυσικό αέριο, ε, ρωσικό και νορβηγικό. Ακόμα δύο σταθμοί ανεφοδιασμού που επιτρέπουν όμως τον ανεφοδιασμό σε υγρό φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το φυσικό αέριο που προέρχεται από το Κατάρ είναι πολύ καλό. Εμείς λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση νη μείον ένα. Νη είναι οι πηγές, μείον ένας που είναι η Λιβύη. Νη μείον δύο θα ήταν κρίσιμη κατάσταση αν ήμασταν, κυρίως σε περίοδο χειμώνα. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρο το, το σύστημα και γι' αυτό και παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης στην Αλγερία και στην Τινησία, ελπίζοντας ότι δεν θα ξεσπάσουν αναταραχές και ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία ε, και προβλήματα. Και για την υπόλοιπη βέβαια Ευρώπη η Ιταλική αγορά παρουσιάζει ε, σημαντικές λαβές όσον αφορά το τι θα πρέπει να γίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη για να βελτιωθεί η ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Από την Ιταλική περίπτωση προκύπτει ότι υπάρχουν δύο σημεία κλειδιά. Τα μακροπρόθεσμα, οι συμβάσεις και οι υποδομές. Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο. Αυτές οι συμβάσεις take or pay τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολλής λόγος για το κύμα, το γεγονό γεγονότων από το 2008 βλέπει και διανύει η βιομηχανία του φυσικού αερίου και η αγορά του φυσικού αερίου. Παλιότερα ήταν προβλέψιμη και βαρετή η αγορά του φυσικού αερίου. Η κατανάλωση του αερίου ανέβαινε κάθε χρόνο κατά 2-3% και το φυσικό αέριο το αγοράζαμε σχεδόν αποκλειστικά με μακροπρόθεμες συμβάσεις, μακροχρόνιες συμβάσεις που συνδέονταν με την αγορά κατέργας του πετρελαίου. Εν τω μεταξύ όμως η ΕΠΑ εξοπλίζονταν για να διαχειριστούν την προβλεπόμενη τους μετατροπή σε μέγα εισαγωγέα ε, φυσικού αερίου. Μόνο την περίοδο 2008, 2000 με 2008 υποβλήθηκαν ε, προγράμματα για 47 εγκαταστάσεις ε, επαναεροποίησης. Από το 2008 όμως άλλαξαν τα πάντα. Στη ΣΥΠΑ η αγορά τελείως ανατράπηκε από το φυσικό αέριο που σχισταολιθώ και έχει καλύψει αυτή τη στιγμή το 78% της εσωτερικής παραγωγής. Το 2010 καμία εισαγωγή πρόσθετη φυσικού αερίου, υγρού φυσικού αερίου, υγροποιημένου μάλλον, δεν ήταν απαραίτητη πια. Οπότε παρέμενα να χρησιμοποιείτε στις τεράστιες ποσότητες ε, ε, ε, εντωμεταξύ οι νέες εγκαταστάσεις, του φυσικού αερίου που έχουν κατασκευαστεί κυρίως στην Αφρική για να εξυπηρετήσουν ε, κυρίως στην Αμερική σε χώρες όπως η Αγγόλα, η Νιγηρία, το Κονγκό βρέθηκαν χωρίς διέξοδο για το αέριό τους που πλημμύρισε την ευρωπαϊκή αγορά και την ασιατική αγορά. Ακριβώς ε, αυτό συνέβαινε ενώ ε, η ζήτηση από ευρωπαϊκής πλευράς έπεφτε ε, λόγω της κρίσης. 6% πτώση είδε η αγορά φυσικού αέριου στην Ευρώπη το 2009 και όλα αυτά οδήγησαν σε μια πόλια όγκων φυσικού αερίου 30 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αντιστοιχούν, για να σας δώσω μια ιδέα, στο σύνολο της κατανάλωσης της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας. Η κατάρρευση της ζήτησης λόγω της κρίσης και η υπερβολική προσφορά λόγω αυτού του, φυσικού, του υγροπημένου φυσικού αερίου που δεν ήθελε πια η Αμερικανική αγορά και που κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη έκαναν ε, να πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου που ονομάζεται spot, αυτό που δηλαδή δεν ε, συνδέεται με τις μακροχρόνιες συμβάσεις. Το 2010 που ήταν η πιο, η ξία στιγμή αυτής της ε, μεγάλης αλλαγής στις τιμές με το, το, το φυσικό αέριο σποτ ε, ε, πολίτο σε μια τιμή 25 δολαρίων. Δηλαδή λιγότερο από το 1 τρίτο του πετρελαίου. Είναι προφανές ότι όλα αυτά τίναξαν τους λογαριασμούς στον αέρα και χρειάστηκε να γίνει νέα διαπραγμάτευση των συμβάσεων ε, των μακροχρόνιων. Αλλά Αμφισβητήθηκε επίσης και η ίδια η χρησιμότητα των μακροχρόνιων συμβάσεων και μιλώ για αυτές τις ίδιες συμβάσεις που αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε την κρίση <clears throat> της ελλειπούς παροχής από πλευράς της Λιβύης. Μετά από λίγους μήνες όμως αλλάζει και πάλι το σενάριο αναφοράς. Βγαίνουμε από την κρίση στην Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να αυξάνεται πάλι η ζήτηση του φυσικού αερίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο όλο ένα και περισσότερες χώρες μεταξύ των οποίων και η Κίνα βασίζονται όλο ένα και περισσότερο στο φυσικό αέριο. Με τα τελευταία σενάρια που έχει επεξεργαστεί η ΙΕΑ προβλέπεται ότι η Κίνα μέχρι το 2035 θα μετατραπεί από μια αγορά όπω η Ιταλική, δηλαδή 90 δις το χρόνο, ε, κυβικών μέτρων ε, το χρόνο, θα μετατραπεί σε μια αγορά που αντιστοιχεί στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, δηλαδή 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μετά υπήρξε η πυρηνική, το πυρηνικό ατύχημα της Ιαπωνίας. Κλείσανε μερικά πυρηνικά εργοστάσια. Λιγότερη πυρηνική πυρηνικά εργοστάσια σημαίνει περισσότερη χρήση φυσικού αερίου και άρα περισσότερη εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου σε αυτές τις χώρες. Φανταστείτε ότι η Ιαπωνία έχει, ένα, έχει 100 σταθμούς επαναεροποίησης, γιατί όλο το φυσικό αέριο που εισάγεται εκεί εισάγεται σε υγρή μορφή. Αν δούμε δε τους φιλόδοξους στόχους ε, περικοπής των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αυτό είναι πολύ θετικό. Θετικά λοιπόν τα νέα όσον αφορά το φυσικό αέριο, όσον αφορά την προσφορά, η βασική καινοτομία είναι ε, το αέριο από σχιστόλιθο. Αλλά σε αυτό υπάρχουν και προβλήματα και ανησυχίες, κυρίως περιβαλλοντικού τύπου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία, για παράδειγμα, είχε απαγορεύσει την παραγωγή του, ενώ η Αγγλία πριν από δύο εβδομάδες ε, δυσκολεύτηκε να απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα παρόμοιο. Φυσικά είναι, αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο αβεβαιότητας ε, και αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα όσα θεωρούνταν δεδομένα μετά το 2008, δηλαδή ένα σωρό φυσικό αέριο και σε καλές τιμές δεν είναι πλέον δεδομένο και γι' αυτό και η Ευρώπη θα πρέπει να ε, αποκτήσει μέσα που θα εγγυηθούν τον ανεφοδιασμό της στο μέλλον. Μέσα σε αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις οι μακροχρόνιες γιατί συνδέουν την Ευρώπη με τους παραγωγούς για πολλά χρόνια διατηρώντας ε, τους συμβατικούς όγκους και προστατεύοντάς τους από την ανταγωνισμό με άλλες περιοχές του κόσμου που διψούν όλα ένα και περισσότερο για φυσικό αέριο. Ας πούμε, τα, τις συμβάσεις με την Gazprom θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η Gazprom την ε, προσεγγίζουν οι Ασιάτες, δηλαδή Κίνα και η Ιαπωνία, που στρέφονται προς την Κασπρόμ για να πάρουν το φυσικό αέριο. Πάλι καλά δηλαδή που έχουμε αυτές τις μακροχρόνιες συμβάσεις που μας εγγυώνται την πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο πόρο ενέργειας. Η εξίσωση είναι απλή. Οι υποδομές απαιτούν επενδύσεις. Και εδώ έρχομαι στο θέμα των υποδομών. Η οι επενδύσει ε, χρειάζονται ε, εταιρείε έτοιμε να αναλάβουν ε, κινδύνους, να αναλάβουν ρίσκα και τα ρίσκα καλύπτονται μόνο με τα μακροχρόνια σε συμβάσεις. Κανείς δεν δεσμεύεται άμα δεν έχει εξασφαλιστεί μέσω αυτών των μακροχρόνιων συμβάσεων. Εξάλλου, οι μεταφορείς που είναι αυτοί που κατασκευάζουν τα αγωγού αγωγούς θα πρέπει να εξασφαλίσουν την πώληση του φυσικού του αερίου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτοί που παράγουν το φυσικό αέριο πρέπει να κάνουν μεγάλες επενδύσεις και για να κάνουν μεγάλες επενδύσεις θέλουν να είναι βέβαιοι ότι θα μπορέσουν και να το πουλήσουν. Αυτοί που κατασκευάζουν τις υποδομές για να μεταφέρουν το φυσικό αέριο και αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα μπορέσουν να τους γεμίσουν τους αγωγούς με φυσικό αέριο. Άρα πάλι μακροχρόνιες συμβάσεις και όσοι αγοράζουν το φυσικό αέριο θα πρέπει να είναι βέβαιοι για μια μακρά περίοδο ότι το φυσικό τους αέριο θα φτάνει μέχρι σε αυτούς μέχρι τον, μέσω των υποδομών. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει πολλά ως Ευρώπη για να διαφοροποιήσουμε τους γεωγραφικούς πόρους ανεφοδιασμού. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό κίνδυνος που συνδέεται με τη διέλευση του φυσικού αερίου. Τα όσα έγιναν στην Τινησία πέρα από την πολύ γνωστή κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πέρα λοιπόν από το κίνδυνο των χωρών παραγωγών, προστίθεται και το κίνδυνο των χωρών που διανύουν η αγωγή, διανύει το φυσικό αέριο πριν φτάσει σε εμάς δείτε τον Nord Stream και τον South Stream και τα δύο αυτά προγράμματα στόχο έχουν να ε, οδηγήσουν το, ρωσικό φυσικό αέριο άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βόρειος ε, αγωγός στην Γερμανία κατευθείαν, ο νότιο κατευθείαν στην Βουλγαρία, χωρίς να διανύουν χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο θέμα των υποδομών έχουμε εμεί ε, ένα τρόπο για να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό για θα πρέπει δηλαδή να στοχεύσουμε με πεποίθηση σε μια πραγματική διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου εσωτερικών, των εσωτερικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέσω μηχανισμών reverse flow μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο από εκεί που υπάρχει, εκεί που χρειάζεται. Και αυτό για να αυξήσουμε την, την ε, ασφάλεια των εφοδιασμών, αλλά και για να έχουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά από ε, άποψη φυσική, πραγματική και εμπορική η διασύνδεση θα επέτρεπε και την βέλτιστη διαχείριση των υποδομών αποθήκευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος του συστήματος. Λόγω της ανεπάρκειας των εσωτερικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του επαναεροποιητή της Ευρώπης, δηλαδή της ισπανικής αγοράς που έχει 7 εγκαταστάσεις επαναεροποίησης. Ε, υπάρχουν ακόμα χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο το ευρωπαϊκό και εξαρτώνται αποκλειστικά από τη Ρωσία για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Για να σας δώσω μια ιδέα για το δυναμικό της διασύνδεσης, δηλαδή μπορούσαμε να φανταστούμε μια Ευρώπη απόλυτα διασυνδεμένη που μπορεί να μεταφέρει κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς προβλήματα, αν λοιπόν γινόταν κάτι τέτοιο, η, ζή, η ζήτηση του φυσικού αερίου θα μπορούσε να καλυφθεί ακόμα κι αν κόβονταν οι εισαγωγές από τη Ρωσία που είναι ο βασικός μας προμηθευτής φυσικού αερίου. Φυσικά αυτό είναι μια πρόκληση που πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στην ουσία πιστεύω χωρίς το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά το να μετατρέψουμε τις 27 ευάλωτες αγορές φυσικού αερίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια μόνη ενιαία αντιαγωνιστική και ασφαλή αγορά είναι ένα ασφαλές πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την ακρίβεια και για την ακρίβεια και, με την, και για την εμπεριστατωμένη σας παρουσίαση. Εγώ δεν θέλω να κάνω σχόλια, μόνο μια πολύ σύντομη ερώτηση θέλω να κάνω για να έχουμε περισσότερο χώρο για συζήτηση. Μια σύντομη ερώτηση που κάπως την απαντήσατε μέσα στα όσα ήδη μας είπατε, κύριε Σκαρόνε. Η πυρηνική ενέργεια διανύει κρίση λόγω των όσων είπαμε. Δηλαδή μια χώρα όπως η Γερμανία το είχε ήδη πει μετά το Τσερνομπίλ αλλά δεν το είχε κάνει. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει το ίδιο. Πάντως θέλει να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια. Εμείς δυστυχώς στην Ιταλία δεν έχουμε καν μπει στην πυρηνική ενέργεια. Εν περιπτώσει. Όπως έλεγε όμως ο κύριος Καρόνη, λιγότερη πυρηνική ενέργεια σημαίνει περισσότερο φυσικό αέριο. Ναι, είναι αξιόπιστη αυτή η διαδικασία υπό το, φω... υπό το φως των όσων συμβαίνουν και αν ναι, πώς θα συμφιλιώσουμε αυτή την υπόθεση, αυτή την προοπτική με την μείωση των εκπομπών ρήπων γιατί και το φυσικό αέριο λιγότερο εκπέμπει από το πετρέλαιο αλλά δεν είναι και απολύτως καθαρό. Αρχίζει η συζήτηση. Παρακαλώ, τρία λεπτά αναπαρέμβαση maximum. Η κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για αυτή την ε, εξαιρετική εισήγηση. Εγώ θεωρώ ότι παρά να κάνουμε παρεμβάσεις, καλύτερα είναι να κάνουμε ερωτήσεις. Στην παρέμβασή σας Ήδη το θίξατε αυτό. Και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το να έχουμε μια τόσο ακριβή παρουσίαση για τα όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και στην παγκόσμια αγορά. Όσον αφορά αντίθετα το ρόλο που εμείς μπορούμε να παίξουμε εδώ, ήθελα να ρωτήσω, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το νέο σενάριο για την αγορά του φυσικού αερίου και αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που ορίζεται από το τρίτο πακέτο. Το σχέδιο κοινωνία των δικτύων είναι ακόμα έγκυρο ή έχει μπει στην άκρη. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ γιατί από αυτού δουλεύουμε. Και δεύτερον, οι κανόνες του τρίτου πακέτου για τον εφοδιασμό για μια επιχείρηση όπως η Έννη στη συγκεκριμένη περίπτωση ευνοούν τις επενδύσεις κατά τη γνώμη σας ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σαρτόρη. Το λόγο έχει ο κύριος Αρλάκη. Παρακαλώ, maximum τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ να συγχάρω κι εγώ τα όπως και ο πρόεδρος Αλμπερτίνη, για την ε, πληρότητα και την συνοπτικότητα της εικόνας που μας δώσατε για την ενεργειακή αγορά και για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. που τόσο μας απασχολεί και μας ανησυχεί. Εγώ θεώρησα βρήκα δύο βασικές ε, σκέψεις που πότε φαίνεται είναι αντιφατικές. Ε, από τη μια πλευρά αυτή η διασύνδεση θα εγγυόταν μεγαλύτερη ασφάλεια και, και επάρκεια, καθώς και διαφοροποίηση στους πηγές ενέργειας για την Ευρώπη, καθιστώντας έτσι λιγότερο πιεστική, πιεστικό το θέμα των ε, αγωγών έτσι καθιστώντας λίγο, εκτό, ε, λίγο εκτός θέματος αυτή την ε, αντιπαράθεση μεταξύ του South Stream και του Ναμπούκο. Μπορεί να ήταν και ένα... Ε, ε, ψευδοπρόβλημα και να χρειαζόμαστε και τα δύο για να είμαστε πιο ασφαλείς. Τώρα, αν από την άλλη πλευρά μιλήσουμε για την διασύνδεση και τα δύο, και οι δύο αγωγοί δεν είναι τόσο επίγον να γίνει. Δηλαδή, αν αυξήσουμε την διασύνδεση θα έχουμε περισσότερη ασφάλεια ή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να θεωρήσουμε πως αρκεί το ένα από τα δύο, η διασύνδεση δηλαδή. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που κάπως ξεκαθαρίζεται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Και έπειτα, από ό,τι κατάλαβα, στην πραγματικότητα οι προοπτικές μας για ασφάλεια και ενεργειακή σταθερότητα μέσο και μακροπρόθεσμα φαίνεται πως βελτιώνονται, αυξάνονται. Δεδομένη της κατάστασης των διεθνών αγορών και του περάσματος από την πυρηνική ενέργεια στις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και άρα και στο φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε κύριε Αρλάκη. Έχουν προσθεθεί και άλλες παρεμβάσεις. Δυστυχώς πρέπει να μειώσω στα δύο λεπτά το χρόνο παρέμβασή σας για να μπορέσουμε να τους σας ακούσουμε όλους όσους ζητήσατε το λόγο. Ο κύριος Τούρμες, δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ, κύριε Σκαρόνη. Σίγουρα χρειαζόμαστε αυτές τις διαφορετικές ροές όσον αφορά το φυσικό αέριο, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές δυσκολίες που επηρεάζουν την κατάσταση και εμποδίζουν ε, την διασύνδεση ε, ανάμεσα στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη είναι κάτι το οποίο έχει μπει στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Βλέπουμε βέβαια να γίνεται κάποια πρόοδος. Αν δούμε τα αποτελέσματα όσον αφορά την οδηγία της ασφάλειας εφοδιασμού και τις σχετικές ρυθμίσεις, ε, διαπιστώνουμε ότι πολλά προβλήματα θα λυθούν. Πάντως, ένα ζήτημα που θέλω να θίξω είναι το εξής. Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αν αφήσουμε την πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ τον όγκο φυσικού αερίου. Τα σενάρια τα οποία χρησιμοποιούν πολύ ε, μεγάλο ποσοστό εναλλακτική ενέργειας έχουν σαν αποτέλεσμα Μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων στα κτίρια και προσπαθούμε να έχουμε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η χρήση. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπογραμμίσετε κύριε Σκαρόνη την εξάρτησή μας από τη Ρωσία. Όμως τότε γιατί υποστηρίζετε το South Stream περισσότερο από τον Ναμπούκο. Γιατί για μας ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε ανεξάρτητοι... Ναι, τελειώνω. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε ανεξάρτητοι από τη Ρωσία, ο καλύτερος τρόπος είναι να λειτουργήσει το Ναμπούκο. Οπότε δεν ε, μπαίνετε ο ίδιος σε αντίφαση με τον εαυτό σας όταν λέτε να είμαστε ανεξάρτητοι από τη Ρωσία, αλλά από την άλλη μεριά στηρίζετε το South Stream. να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο σε όλους αν δεν τηρείτε το χρόνο των δύο λεπτών. Προβέρα που είναι Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Σκαρόνη που ήταν πραγματικά πολύ ε, περιστατωμένη η εισήγησή του. Έθιξε πολλά θέματα, ίσως όχι όλα, αλλά πάντως ε, ήταν... Ε, Δύο ερωτήσεις ε, όσον αφορά την έκβαση του δημοψηφίσματος στην Ιταλία που μας απαγορεύει να κάνουμε οποιαδήποτε μελλοντική επιλογή για το ποια θα είναι για, την ενέργεια. Δύο απλούστατες ερωτήσεις. Η γνώμη σας για το μέλλον της Λιβύης όχι για το στρατηγικό και πολιτικό μέλλον, γιατί αυτό φαίνεται νεφελώδες και όλο ένα και χειρότερο. Αλλά η Λιβύη ως ενεργειακός πόρος και κυρίως ο ρόλος που θα της επιφυλαχθεί μετά την αλλαγή της κατάστασης, ο ρόλος της έννοια και της χώρας μας δηλαδή. Ναι. Η ήττα τη πυρηνική ενέργεια θα έπρεπε να αποτελεί τον θρίαμβο για την ε, ανανεώσιμη ενέργεια και θα ήθελα να ξέρω την γνώμη σας, ε, αιτιολογημένη τεχνικά, για τις διαστάσεις, για το μέλλον των εναλλακτικών πόρων και για τις ε, συγκεκριμένες διαστάσεις αυτού του μέλλοντο στην καθημερινή ζωή και στην ποιότητα ζωή των πολιτών μα. Σα ευχαριστούμε κύριε Προβέρα. Το λόγο έχει ο κύριος Ντεάντζελης. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ εκτίμησα ιδιαίτερα την έκθεση του κ. Σκαρόνη. Πολύ ακριβής. Και πλήρης. Και, κυρίως ε, έχω να κάνω δύο ερωτήσεις για να μην χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Εγώ έχω κάπως διαφορετική άποψη, με την έννοια ότι πιστεύω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν ε, ξεκινήσαμε ποτέ με την πυρηνική ενέργεια στην Ιταλία, εννοεί ο μιλητής. Και ο προβληματισμός που κάνω και με βάση τα όσα συνέβησαν τελευταία είναι μήπως θα έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο και με μεγαλύτερο θάρρος και πεποίθηση στις ανανεώσιμες και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Και με βάση μάλλον με βάση να, να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο μιας υπερβολικής εξάρτησης από τη Ρωσία. Γιατί βλέπω ότι έτσι θα είχαμε ε, μια πιο ελεύθερη αγορά. Πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα της εξάρτησης. Ευχαριστούμε κύριε Ντεάντζελες. Δύο λεπτά στον κύριο Χατζηγεωργίου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον φιλοξενούμενο μας. Υπάρχουν, ε, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για αποθέματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο που ε, οι διοκτήτες τους είναι το Ισραήλ και η Κύπρος. Και ήθελα να ξέρω τι εικόνα υπάρχει γύρω από αυτά τα αποθέματα, ε, ποιες εξελίξεις υπάρχουν και εάν θεωρεί ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βασίσει ένα μέρος ε, της προμήθειάς της ε, σε αυτά τα αποθέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηγεωργίου. Ριέρα Μαντουρέλ για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον συγητή μας ε, εδώ, τον κύριο Σκαρόνη. Και θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς που θα πάρουν στη συνέχεια το λόγο για τη συμμετοχή τους στην ακρόαση αυτή. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Πρόεδρος, Υπάρχει ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ και τις δύο επιτροπές μας. Πρόκειται για την ενέργεια. Γι' αυτό και οι δύο πρόεδροι ε, οργάνωσαν από κοινού την ακρόαση αυτή. Ε, συμφωνούμε με πολλές από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν ήδη οι συνέδρεφοι και με τα σχόλιά τους όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Θα περιμένω βέβαια και τους άλλους εισηγητές να δω ότι θα πούνε και εκείνοι, γιατί και για αυτούς θα έχω σίγουρα διάφορες ερωτήσεις, αλλά στους ακούσω προηγουμένως, μήπως έχουν ε, ε, συμπεριλάβει στις εισηγήσεις τους τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Πάντως, Μία πρόταση θα ήταν οι δύο εισηγητέ οι επόμενοι να παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους και μετά να συζητήσουμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε καλύτερα τις ερωτήσεις μας. Τώρα, τι θέλω να ρωτήσω και έχω και να σχολιάσω λίγο για τη δουλειά μας εδώ. Η ενέργεια για διάφορες περιοχές στον κόσμο αποτελεί ένα στοιχείο ολοκλήρωσης μερικές φορές και βοηθάει και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Οπότε είναι λογικό το ίδιο να συμβεί και στην νότια πλευρά της Μεσογείου. Η ασφάλεια, η σταθερότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η δικιά μας ενεργειακή ασφάλεια απειλείται εφόσον δεν υπάρχει ασφάλεια από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς να κάνουμε όταν ετοιμάσουμε διακόπτει ο πρόεδρος. Έχετε ξεπεράσει κατά 50% το χρόνο σας. Λυπάμαι, γι' αυτό σας διακόπτω. Συνιάσκη, δύο λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω όμως. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακούσαμε για την ε, ασφάλεια του ε, ανεφοδιασμού και για τις ε, μακροπρόθεσμες ε, συμβάσεις και τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει της Gazprom, ε, τους αγωγούς North Stream και South Stream. Αυτά οδηγούν σε σημαντική διαφοροποίηση στην κεντρική και ε, ανατολική Ευρώπη. Εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από την Gazprom. Οι χώρες αυτές είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν έχουν πρόσβαση στον, στους αγωγούς South Stream και North Stream. Εξάλλου υπάρχουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις με την Gazprom. Οι χώρες αυτές ε, δεν ε, λαμβάνουν καμία ε, στήριξη όμως. Και οι αγωγοί αυτοί έχουν εξαιρεθεί από το τρίτο πακέτο, γι' αυτό ερωτούμε πώς θα διασφαλιστεί ο ανεφοδιασμός στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Θέλουμε η Κάσπρομ να μην ε, έχει μονοπόλιο στην ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η μακροπρόθεσμες ε, συμβάσεις δίνουν ασφάλεια κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις διότι μπορούν έτσι να βασίζονται σε αυτές. Δεν, ξέρω, όμως ε, εάν είναι ε, χρήσιμες οι συμβάσεις αυτές για τους καταναλωτές, διότι ε, εμφανίζονται νέες πηγές ενέργειας, ενέργειας όπως είναι το αέριο από και οι μακροπρόθεσμες αυτές συμβάσεις θα δυσκολεύσουν την διαφοροποίηση των τιμών και των προϊόντων. Ε, επίσης, όταν μιλάμε για ε, διαφοροποίηση, εσείς μιλήσατε για το Nord Stream και το South Stream, αλλά αυτό δεν είναι ε, διαφοροποίηση. Πάλι μιλάμε για ρωσικό αέριο και δεν αναφερθήκατε στον Ναμπούκο. Αυτό τουλάχιστον θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο χθε ε, η Herald Tribune ε, έγραφε στην ε, πρώτη σελίδα ότι ο αγωγός South είναι μια μεγάλη μπλόφα που απλά θέλει να εξασθενήσει το πρόγραμμα Ναμπούκο. Δεν ξέρω τι γνώμη θα είχατε εσείς για το άρθρο αυτό και... Τρίτον, τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσει όσον αφορά την ε, ανασφάλεια που προκαλείται από τους προμηθευτές μας. Αναφερθήκατε στην Βόρεια Αφρική, ε, βλέπουμε ποια είναι η πολιτική κατάσταση αυτή. Μπορεί όμως να αντιμετωπίσουμε το ίδιο με τη Ρωσία. Σύντομα θα ασχοληθούμε με την έκθεση ε, εξωτερικής διάστασης της ενέργειας που θα λαμβάνει υπόψη και άλλες ε, χώρες. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, ποια μέσα ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Εσείς τι γνώμη έχετε για την πρόταση του Προέδρου και για την κοινή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σκαρόνη για την παρουσίασή του. Το επόμενο εξάμεινο, κύριε Σκαρόνη, θα είναι το εξάμεινο της μάχης των αγωγών, από ό,τι φαίνεται, για να αποφασίσουμε σε ποιον αγωγό θα καταλήξουμε. Η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν, εδώ και μία εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι θα επιλέξει έναν αγωγό, τον οποίον θα προμηθεύει από όλους τους επίδοξους αγωγούς που συζητάμε. Η ερώτησή μου ως προς το θέμα των αγωγών είναι διαφαίνεται κατά τη γνώμη σας μία συγχώνευση των υποσυζήτηση αγωγών. Γιατί ο κύριος προμηθευτής είναι το Σαχντενής του Αζερβαϊτζάν με 16-17 δισεκατομμύρια cubic ε, meters εφοδιασμό. Άρα αν διασπαστεί στις εταιρείε δεν μπορεί να προμηθεύσει τελικά κανέναν. Η δεύτερη τοποθέτησή μου είναι για τον νότιο ε, διάδρομο. Πώς βλέπετε το ρόλο, πώς βλέπετε το ρόλο, πώς βλέπετε το ρόλο των Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, στον εφοδιασμό με γκάς του νοτίου διαδρόμου. Αν θεωρείτε κλειδί την επίλυση του θέματος του πολιτικού με το Ιράν, το οποίο κατά τη γνώμη μου αν επιληθεί θα αλλάξει όλο τον οικονομικό και ενεργειακό χάρτη στο νότιο και βόρειο κομμάτι της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζαβόλ. Τζαβέλα, Μίλαν μόνο δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον κύριο Σκαρόνι για την παρέμβασή του. Δεν ξέρω τώρα αν δεν κατάλαβα καλά. Πάντως δεν άκουσα δεν κατάλαβα για την άποψή του όσον αφορά την ενέργεια από μη συμβατικέ πηγέ. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ ε, όσον αφορά την ενέργεια από σχιστόλθε στι ΗΠΑ, για παράδειγμα. Η Πολωνία έχει μεγάλε εξαγωγέ τέτοιε. Οπότε, να ρωτήσω και όπω και η κυρία Κολάσκα, και εγώ διάβασα τη Herald Tribune χτε στην πρώτη σελίδα το άρθρο που έλεγε ότι το South Stream με τον Ναμπούκο βρίσκονται σε αντιπαράθεση παρόλο που και τα δύο είναι κάτι εικονικό και λίγο ρεαλιστικό. Ποιο είναι ο στόχο τη ακρόαση αυτή, είναι ακριβώ να καταλάβουμε. Λοιπόν, για πείτε μα εσεί όσον αφορά τι διάφορες πολιτικές που κυκλοφορούν, τι προβλέπουν όσον αφορά τον εφοδιασμό από την Νότια Μεσόγειο, τι θα γίνει με τον εφοδιασμό αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μιλανμόν. Ο κύριος Ράνστορφ, δύο λεπτά παρακαλώ. Grazie Presidente, grazie Relatore Scaroni. Ε, una, una domanda molto corta. Che Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνας για τα βορειοαφρικανικά προγράμματα, τα ενεργειακά. Ευχαριστώ. Μας κάνατε να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Κύριος Μετζάνος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκαρόνη ε, για την ε, ερώτησή του. Ευχαριστώ που προσπαθείτε να μειώσετε την εξάρτησή μας από την ε, Ρωσία. Η δική μου πατρίδα, η Σλοβακία, εξαρτάται κατά 100% από το ρωσικό αέριο. Είναι όμως αβέβαιο το μέλλον του σχεδίου αυτού μία ερώτηση ε, σχετικά με τα αποτελέσματα του Ιταλικού Δημοψηφίσματος ε, για ε, για το, την πυρηνική ενέργεια. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον ε, της Ευρώπης. Ε, θα μπορέσουμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Και πώς θα πετύχουμε στον αγώνα μας κατά της αλλαγής του κλίματος και πώς βλέπετε εσείς τις νέες ασιατικές τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Κυρία Τικάου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η σχέση Μεσογείου και Εύξηνου Πόντου. από στρατηγικής πλευράς, διότι ο Εύξηνο Πόντος είναι το, πέρασμα για την ε, Κασπία ε, θάλασσα. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντική η Μεσόγειος ε, για την ε, ασφάλεια αναφοδιασμού στην Ευρώπη και γι' αυτό θεωρούμε τον αγωγό Ναμπούκο και, την, και τον αγωγό της Αδριατικής, τον σύνδεσμο Αζερβαϊτζάν, Τουρκίας και Ευρώπης, όλοι ε, όλες αυτές οι διαδρομές είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια αναφοδιασμού στην Ευρώπη. Ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς βλέπετε το πρόγραμμα TEC. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει έτσι να διασφαλιστεί ε, η απαραίτητη ενέργεια μέσω της Βορειοαφρικής. Και όσον αφορά το πακέτο προστασ... καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Ε, πώς το βλέπετε αυτό, ευχαριστώ. Ηλα... Πρόεδρος. Έχουμε και τον κύριο Βονουά που είναι ένας από τους ε, ομιλητές μας, αλλά θέλει και αυτός να ρωτήσει κάτι τον συνάδελφο. Οπότε θα ακούσουμε και τον κύριο Βινουά. Παρακαλώ κύριο Βινουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σκαρόνη και εγώ για τόσα είπε. Αναφερθήκατε στις ε, μακρόχρονες συμβάσεις. Εσείς πώς βλέπετε το περιθώριο ελαστικότητας που έχουμε για να βελτιώσουμε το σύστημα. Υπάρχουν ε, οι αγορές spot, όπως είπαμε πριν, για σας πρέπει να μειωθεί η διάρκεια τέτοιων μακροχρόνιων συμβάσεων, πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστώ που ήσασταν και συνεκτικός και σύντομος. Πολλές ερωτήσεις. Και ο εισηγητής μας σίγουρα θα μπορέσει να συμπυκνώσει τις απαντήσεις του σε 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα θέματα που θίξατε. Πρώτα απ' όλα. Πολλοί από εσά ρώτησαν το ίδιο πράγμα και αναφέρθηκε χτες στην Herald Tribune. Ναμπούκο εναντίον South Stream. Δεν είναι σε αντίθεση όμως αυτά τα δύο, γιατί South Stream είναι Ρωσία, Ναμπούκο είναι Ουκρανία. Οπότε δεν υπάρχει εκεί πρόβλημα. Με τον Ναμπούκο θα έχουμε εξαγωγές από το Τουρκμενιστάν, Ιράκ και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του Ναμπούκο. Είμαστε αυτοί που έχουμε οικοδομήσει το μεγαλύτερο μέρος αγωγών, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον και ποτέ δεν είδαμε να υπάρχει άλλος ε, αγωγός ε, που να έχει χρειαστεί τόσα χρήματα. Για μας δεν πρόκειται για ένα στέρεο σχεδιασμό. Αν θέλετε, αυτή είναι, αυτός είναι ο δικός μας συλλογισμός. Είναι δύσκολο όταν στην ανάπτυξη ενός αγωγού δεν έχουμε τον παραγωγό. Πάντως δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο αγωγούς. Τώρα, το έρωπο σχιστόλιθο. Εμείς είμαστε η ευρωπαϊκή επιχείρηση που έχει εμπλεχτεί περισσότερο. Ήδη στις ΗΠΑ παράγουμε τέτοια ενέργεια. Ε, και στην Πολωνία προσπαθούμε ε, επίση να προχωρήσουμε στην Ουκρανία, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι είναι δύο πολλά υποσχόμενε χώρε για το αέριο αυτό. Ε, δεν το έχουμε ακόμα βρει, είμαστε ακόμα στη φάση των ελπίδων και όχι στη φάση της πραγματικότητας. Να σας πω ότι έχουμε επίσης συμμετοχή για το αέριο που σχιστόλουθα στην Κίνα, στην Ισία και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Δημοκρατία στη Βόρεια Αφρική, βεβαίως. Οι μεταβατικές περίοδοι είναι πάντοτε δύσκολες. Όλοι προτιμούν να έχουν τον ίδιο συνομιλητή για πάντα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι θα περάσουμε μια δύσκολη περίοδο και σίγουρα ότι προτιμάμε να έχουμε να κάνουμε με δημοκρατικές χώρες παρά να έχουμε να κάνουμε με τύραννους. Δεκτάτορες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ε, υπομένουμε αυτή την περίοδο, την περίπλοκη, αλλά είμαστε υπέρ φυσικά της ε, δημοκρατίας στη Βόρεια Αφρική. Δύο λόγια για το θέμα ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο κτλ. Και εγώ πιστεύω πως η χρυσή περίοδο του φυσικού αερίου θα διαρκέσει ίσως 15 χρόνια και ίσως έπειτα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταφέρουν να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντικαταστήσουν τους υδρογονάνθρακες γιατί όχι και το φυσικό αέριο. Σίγουρα η σημερινή κατάσταση με τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας μας δείχνουν ότι οι ανανεώσιμες είναι πολύ ε, ακριβές. Ας πούμε η φωτοβολταϊκή στην Ιταλία κοστίζει έξι φορές παραπάνω από τη θερμική ενέργεια και το πληρώνει ο καταναλωτής γιατί στην Ιταλία πάει στην ε, τιμή του, της θέρμασης αλλά σίγουρα είναι όταν το, το, το, το χρειαζόμαστε είναι θέμα δηλαδή αποθήκευση και όχι ισορροπίας του, και, ισορροπία του δικτύου που δεν το έχουμε ακόμα λύσει. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια είναι το μέλλον, αλλά είναι ένα μέλλον επί το οποίο πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες. Γιατί οι σημερινέ ανανεώσιμε, αυτέ που ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμή, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στι απαιτήσει ε, των καταναλωτών μα. Πρέπει δύο λόγια, δεν θυμάμαι ποιο, αλλά για αυτό που εγώ ονομάζω την ε, λεκάνη του Λεβάντε, ανάμεσα στην Κύπρο, στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Εκεί δεν είναι απλώς ε, κάτι που υποψιαζόμαστε, είναι ένα τεράστιο κοίτασμα, θαλάσσιο κοίτασμα, τεράστιο ε, ανοιχτή θάλασσα που λέμε δηλαδή. Ήδη το Ισραήλ το εκμεταλλεύεται και παράγει 20.000 βαρέλια την ημέρα. Εμείς εντάξει μιλάμε για βαρέλια και για το φυσικό αέριο για να έχουμε την ίδια μονάδα μέτρησης που είναι μια σημαντική ποσότητα και που επιτρέπει στο Ισραήλ να ξεπερνά εν μέρη μάλλον να συμπληρώνει την υπόλοιπη ροή που έρχεται από την Αίγυπτο. Βέβαια θα είναι ε, δαπανηρόβο το φυσικό αέριο γιατί είναι βαθιά στη θάλασσα μέσα, αλλά σίγουρα αποτελεί την πηγή του μέλλοντος για κάποια χρόνια. Το Κατάρ κάποιο το ανέφερε. Είναι μεγάλος παραγωγός βέβαια και ο μεγαλύτερος παραγωγός υγρού ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου και έρχεται εδώ στην Ευρώπη και εμείς οι ίδιοι το εισάγουμε. Και έχει αυτό το κοίτασμα που ονομάζεται South Pass και που είναι μοιρασμένο στα δύο ανάμεσα στο Κατάρ και το Ιράν. Φυσικά το Ιράν δεδομένων των ε, ε, κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί το δικό του κομμάτι του κοιτάζοντας, αλλά μία μέρα των ημερών, όταν θα προβληθούν τα προβλήματα εύχομαι αυτό να γίνει ε, μέσα στο εγγύς μέλλον θα έχουμε ακόμα μια πηγή ε, ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Επίσης άκουσα να γίνεται λόγος για ανεφοδισμό από τη Ρωσία, τη Σλοβακία που εξαρτάται 100% από τη Ρωσία. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ακριβώ γι' αυτό μιλώ για ευρωπαϊκή διασύνδεση, διεκτίωση. Πρέπει δηλαδή επειδή κάποιο Σλοβάκο βουλευτή μίλησε, γι' αυτό τη φέρω σε παράδειγμα. Ναι, εντάξει, προμηθεύεται από τη Ρωσία, αλλά σε περίπτωση ανάγκη να έχει του αγωγού που τη επιτρέπουν να εισάγει αέριο που έρχεται από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία. Δηλαδή, αν η Σλοβακία ήταν διασυνδεδεμένη και με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε περίπτωση ατυχήματο ή της νιωστής ε, αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, να μην μας νοιάζει, να, μην, να, χρειάζεται, να μπορεί να πάρει από τι άλλε χώρε. Αλλά επειδή δεν ισχύει αυτό σήμερα, δεν έχουν γίνει απαραίτητε διασυνδέσεις στην Ευρώπη, δεν μπορούμε και να μεταφέρουμε φυσικό αέριο από τη μια χώρα της Ευρώπης στην άλλη. Και όταν μια χώρα αντιμετωπίζει επίγουσα ανάγκη, μένει μόνη της. Το είδαμε πριν από 1,5 χρόνο τη Βουλγαρία, τη Σλοβανία. Μέσα στο κρύο, φουλ χειμώνα και τα νοσοκομεία ήταν παγωμένα. Και δεν μπορούσαμε να τους πάμε το αέριο. Παρότι η Δυτική Ευρώπη έπλεε στο αέριο αλλά δεν υπήρχαν υποδομέ για να μην γίνει η μεταφορά αυτή από την Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική. Αυτή είναι η ιδέα που θέλω να σας μεταδώσω. Να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Αρχή για το φυσικό αέριο, που να είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση εντός της Ευρώπης, όπως το κάνουν και στη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ, από το ένα, ε, μια πολιτεία στην άλλη πάει ελεύθερα το φυσικό αέριο. Πολύ ανταγωνιστική αγορά. Και έτσι λύνεται και το πρόβλημα. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάπω απαλύνεται το, το πρόβλημα της ασφάλειας ανεφοδιασμού. Τώρα, για τι μακροχρόνιε συμβάσεις. Αυτές τι take or pay. Που όχι μόνο εμεί οι Έννοι, αλλά και οι Gas de France, οι Aeon, έχουν τέτοιου είδου μακροχρόνιε συμβάσει με του παραδοσιακού προμηθευτέ φυσικού αερίου Νορβηγία, Ρωσία, Αλγερία, Λιβύη. Αυτές οι συμβάσεις λοιπόν αυτή τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές SPOT που συνδέονται με τη τιμή του πετρελαίου αυτές τις αναδιαπραγματευόμαστε με τώρα. Είτε δηλαδή αν και διατηρήσουμε το μηχανισμό που τα συνδέει με το αργό πετρέλαιο τις τους μειώνουμε για να ανταγωνιστούν το gas spot, είτε αν διατηρήσουμε τις μακροχρόνιες συμβάσεις, δηλαδή αγορά και πώληση μακροπρόθεσμα, συνδέουμε τις τιμές με την αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή στο National Balancing Point, που είναι η αγγλική, η βρετανική αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι η αγορά όπου καθημερινά συναλλασσόμαστε σε μεγάλους όγκους φυσικού αερίου. Μπορούμε να συνδέσουμε δηλαδή ε, την παροχή σε αυτή την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναφέρονται οι αγορές ε, σε όλες τις εφημερίδες είναι δηλαδή ένα σίγουρο σημείο αναφοράς. Κίνα και Βόρειο Αφρική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρουσία κινέζικη στην Βόρεια Αφρική. Υπάρχει στους υδρογονάνθρακες η κινέζικη παρουσία στην ε, Αφρική νοτίως της Σαχάρας, όχι όμως στη Βόρεια Αφρική. Πώς είπατε, Α, ναι, ναι, η ερώτησή σας για τη Λιβύη. Εξαίρεση της αποκλεισμός της Λιβύης. Υπάρχει κινέζικη παρουσία στη Λιβύη. Όχι, δεν υπάρχει ή και αν υπάρχει είναι ασήμαντη εντελώ. αμεληταία. Δεν είναι παρούσα η Κίνα στη Βόρεια Αφρική. Και έτσι νομίζω πως απάντησα σε όλα. Ξέχασα κάποιον. Κυρία Τζαβέλα, Κάποια διευκρίνηση θέλετε, παρακαλώ. Τα συγχώνευσης, την πιθανότητα συγχώνευσης των αγωγών μετά την απόφαση του Αζερβαϊτζάν να προμηθεύσει έναν αγωγό. Πώς τη βλέπετε. Α, ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ναι, στην πράξη το Αζερβαϊτζάν είναι ο, ο αποκλειστικό προμηθευτή του Ναμπούκο. το, ο Ναμπούκο θα αρχίσει να λειτουργεί αν το φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊζάν τουλάχιστον 15 δις κυβικών μέτρων δοθεί στο κονσόρτσιο του Ναμπούκο. Τώρα δεν ξέρω αν οι όσοι συμμετέχουν εκεί πέρα θα ξεκινησουν δαπανωντας δαπανώντα 10-12 δις ευρώ μόνο για μια σύμβαση. Γιατί εγω εγώ κατασκευάσω ένα αναγωγό, δαπανίσω 10-12 δις ευρώ και μετά δεν έχω παροχή, δεν έχω αντιστάθμα, δεν έχω απόδοση θα προτιμούσα να, δώσω, να τα δώσω στην κατασκευή του αγωγού και νομίζω πως αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αλλά κοιτάξτε, μιλάει για κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν γιατί εμείς δεν είμαστε εμ, συνεταίροι στον Ναμπούκο. Κάποιος ακόμη δεν το λόγο. Ευχαριστώ. Πώς βλέπετε κύριε Σκαρόνη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία, το όχι δηλαδή στην πυρηνική ενέργεια. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, οι Ιταλοί έχουν πολύ δύσκολη σχέση με την πυρηνική ενέργεια εδώ και χρόνια. Και με τους αποτεφρωτές έχουν πρόβλημα, με τις νέους αυτοκινητόδρομους, με τους σιδηρόδρομους. Κάθε δηλαδή δημόσιο έργο το οποίο κάπως ε, είναι έτσι ε, ε, παρεμβατικό τους κάνει να αντιδρούν. Εγώ πιστεύω πως αυτό το δημοψήφισμα θα θάψει την πυρηνική ενέργεια στην Ιταλία για τα επόμενα δέκα χρόνια. Δεν θα ήμουν τόσο βέβαιος για άλλες χώρες, γιατί είναι παράξενο, δεν ξέρω αν το είδατε, χτες η Ιαπωνική κυβέρνηση απόφασε ότι θα προχωρήσει, θα συνεχίσει με την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή η χώρα που έζησε τη Φουκουσίμα συνεχίζει με την πυρηνική ενέργεια. Στον κόσμο υπάρχουν 450 πυρηνικές εγκαταστάσεις, δεν είναι μόνο δύο-τρει. και έχω την εντύπωση ότι καμιά χώρα στον κόσμο δεν έκανε ε, δημοψήφισμα για να αφήσει την πυρηνική ενέργεια. Εμείς ούτε καν είχαμε μπει, οπότε Εν πάση περιπτώσει, αυτέ είναι οι επιλογέ των συμπολιτών μα και δεν τι αμφισβητώ, γιατί ούτω ή άλλω και στην εταιρεία μου δεν ασχολούμαι εγώ με την πυρηνική ενέργεια. Και μάλιστα δήλωσα σε άσχετο στιγμή ότι δεν ήταν ε, δική μα υπόθεση. Άρα δεν νιώθω να με αφορά. Βεβαίω, αν μπορώ να προσθέσω μια λεπτομέρεια αυτό, το οποίο γοητεύει όσου ασχολούνται με την ενέργεια και την πυρηνική ενέργεια είναι ότι ε, ε, δεν έχει εκπομπέ. Επειδή όλοι όσοι παράγουν ενέργεια έχουν πάθει αυτή τη μανία με τις ε, εκπομπές, το να φτιάχνουν ενέργεια ενώ δεν υπάρχουν εκπομπές είναι ένα ονειρεμένο πράγμα. Και γι' αυτό και όλοι εγωιτεύονται και γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη τάση υπέρ της ενέργειας γιατί έχουν ε, μηδενική εκπομπή που είναι, ε, ε, οι είναι ο εχθρό αυτή τη στιγμή. Σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Σκαρόνη για την παρουσίασή σα για την ακρίβεια και την ε, συντομία με την οποία και την περιεκτικότητα με την οποία απαντήσατε στι ερωτήσει μας. Πραγματικά είμαι γεμάτος θαυμασμό για το πώς παρουσιάσατε τη χώρα μας και την τόσο μεγάλη αυτή επιχείρηση. Να σας πω ότι μιλάμε όντως για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρμόδιας αρχής για τη διασύνδεση. Εκεί όπου δεν υπάρχει ποσότητα φυσικού αερίου θα μπορούσε το δίκτυο να αντικαταστήσει αυτή την λήψη και θα μπορούσε να είναι και ενεργειακή εξοικονόμηση αν υπήρχε σύνδεση. Και τώρα θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Ρέλα. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο και από εδώ και μπρος θα προεδρεύσετε εσείς. Μπες περιπτώσει. Θέλεις, αν θέλεις, Έλα να κάτσεις τη θέση σου. Κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα να συνεχίσουμε. Καλύτερο θα ήταν αν και οι δύο προσκεκλημένοι, και οι δύο επόμενοι προσκεκλημένοι, Καλά, θα το κάνουμε ένας-ένας. Ε, θα έρθει εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Φρανσέσκο Δελφροκάσια, που είναι ε, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΑΓΑΣ. Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι παρόμοιο με αυτό που μόλις ακούσαμε. Ε, από τεχνικής αποψή είναι όλα έτοιμα, όχι ακόμα. Ωραία, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Δεν ε, θα ε, μακρηγορήσω κατά την εισαγωγή μου. Θα ακούσω μια δεύτερη γνώμη για το θέμα που σήμερα μας απασχολεί. Ε, χωρίς πολλά λόγια, σας δίνω το λόγο κύριε Τελεφλόρ. Παρακαλώ. Σα ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους σας. Όντως, είμαι από την Εναγκάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε εδώ. Και τους δύο πρόεδρους των δύο επιτροπών που οργανώνουν αυτήν την ακρόαση. Συζητάτε το πακέτο υποδομών αυτήν την εποχή, την εποχή και τίθεται σε εφαρμογή ο τελευταίος κανονισμός σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ασχοληθούμε, όπως λέει και ο τίτλος ακρόασης αυτής, για τις δυνατότητες διασύνθεσης των διαφόρων ενεργειακών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας μιλήσω και για την ασφάλεια εφοδιασμού. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη μας και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη νότια πλευρά της Μεσογείου θα επικεντρωθώ στην παρουσίασή μου για την ε, άποψη έτσι όπως αυτή προκύπτει από την ιβηρική Χερσόνησο, από την οπτική γωνία της ιβηρικής Χερσονήσου. Θα σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα την ε, επιχείρησή μου, την Αναγάς, που είναι διαχειριστής ε, με πλειοψηφία του φυσικού αερίου στην Ισπανία και στην Ιβυρική Χερσόνησο. Έχουμε 10.000 αγωνικά χιλιόμετρα Μιλάμε 72-80 ε, μπαρ πίεση, αγούς δηλαδή υψηλής πίεσης και διαθέτουμε και βασικές υποδομές ολόκληρη την Ισπανία. Έχουμε εγκαταστάσεις και υπόγειες. Η αναγκάς δηλαδή είναι μια επιχείρηση η οποία ε, δουλεύει ε, μέσα στην ρυθμισμένη αγορά της Ιβερικής Χερσονήσου. Είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση ε, ενταγμένη στο χρηματιστήριο, με μετοχές δηλαδή και μετόχους, 75% είναι το free float, ελεύθερη ροή με επενδύσεις που ανήκουν σε διάφορες χώρες του ΟΣΑ. Το υπόλοιπο 25% βρίσκεται στα χέρια διάφορων τοπικών και περιφερειακών ε, επιχειρήσεων, της ΣΕΠΗ, της Oman Oil Corporation και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από διάφορες ανεξάρτητες προσωπικότητες. Αυτή η ανεξαρτησία είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα έλεγα ότι η ΕΝΑΓΑΣ έχει ακολουθήσει μία διαδικασία η οποία την έχει βοηθήσει να δραστηριοποιείται επί 10 χρόνια τώρα με τον ίδιο αυτό τρόπο ανεξάρτητης προσέγγισης. Θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, παρουσιάζοντάς σας επιχειρήματα ή απαντώντας σε επιχειρήματα, το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο καθηγητής Σκαρόνη. Είχαμε μια κρίση που ξεκίνησε από τις αρχές του 2001. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Βινό να χρησιμοποιήσω τον χάρτη αυτό που μας έχει παρουσιάσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχω παρουσιάσει πολλές φορές ε, μέχρι τώρα. Η ερμηνεία βέβαια μπορεί να είναι διαφορετική κάθε φορά. Είχαμε λοιπόν το ξεκίνημα της κρίσης τότε στις αρχές του 2009 που έπληξε και τους εταίρους μας κυρίως τις χώρες που βλέπετε εδώ με κόκκινο. Βρίσκονται περισσότερο στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είχε όμως ε, καμία επίπτωση πάνω στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αντιμετωπίζουμε κι εμείς ε, κάποια προβλήματα το φυσικό αέριο το οποίο μπαίνει στην Ιβυρική Χερσόνησο είτε από τη Βόρεια Αφρική είτε υπό τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου από διάφορες χώρες της Υπήρου δεν μπορεί να περάσει από τα Βόρεια Πυρηναία προς την υπόλοιπη Ευρώπη λόγω προβλημάτων διασύνδεσης. Επίσης, ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει έτσι ώστε να υπάρχει μία κατεύθυνση της ροής από την παραγωγή προς την κατανάλωση. Αλλιώς δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εξαιτία αυτή τη κατάσταση λοιπόν ξεκίνησαν κάποια σχέδια, κάποια προγράμματα ώστε να αλλάξουν υποδομέ και να επιτρέπουν την ροή αυτή προ την αντίθετη κατεύθυνση. Καταρχήν λοιπόν η Βυρική Χερσόνησος είχε εγκαταστάσεις εισαγωγής που εξυπηρετούσαν και τους εταίρους μας εξαιτία της αλληλεγγύης ε, που θέλαμε να ισχύει. Από την 1η Ιανουαρίου του 2009 λοιπόν είχαμε μια διασύνδεση με την Αλγερία που περνούσε από το Μαρόκο, ήταν ε, ο αγωγός ε, Μαρόκο Ευρώπης από το 2006 και όπου η κατασκευή του κράτησε αρκετά χρόνια. Επίσης είχαμε και 7 εγκαταστάσεις επανεροποίησης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Όμως η μεταφορά, η φυσική μεταφορά μέσω των πυρηναίων, όπως σας είπα, η δυνατότητα μεταφοράς ήταν μηδενική εκεί. Εδώ και μερικές εβδομάδες λοιπόν έχουμε έναν αγωγό ο οποίος συνδέει απευθείας την Αλγερία με την Ισπανία. 8 φορές το χρόνο και μπορεί να αυξηθεί η δυνατότητα πολύ περισσότερο αν προσθέσουμε κάποιες επιπλέον υποδομές. Τόσο λοιπόν και το υγροποιημένο αέριο και όσο και το φυσικό αέριο μπορούν να προσφέρουν επιπλέον ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η οικοδόμηση του Μελκάς έχει νόημα εφόσον το δούμε σαν μια νέα διαδρομή. Πολύ περισσότερο από ό,τι σαν μια πηγή απλώ εφοδιασμού τη Ιβηρική Χερσονήσου. Θέλουμε λοιπόν να αποφεληθούμε από αυτό, διότι Καταλαβαίνετε ότι για να οικοδομηθεί ένα αγωγός να φτιαχτεί η υποδομή δηλαδή χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια, άδειε, χρήματα κλπ. Τώρα, όπως είπαμε, η δυνατότητα διασύνδεση ανάμεσα στην Ιβερική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μηδενική. Αρχικά υπήρχε αυτή η μια κατεύθυνση μόνο ροή για να ε, τηρηθούν κάποιε συμβάσει που είχαν γίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη τρει φορέ το χρόνο. Πολλέ ε, φορέ προσπαθήσαμε να αυξηθεί η δυνατότητα παροχή μέσω των Πυρηναίων, όμω ακόμα και παρά τη δήλωση τη Βαρκελόνη του 2005 δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν τοπικέ πρωτοβουλίε παρά μόνο αργότερα. Πολύ αργότερα. Παρόλο που υπάρχει η αλληλεξάρτηση με την Γαλλία και έγιναν προσπάθειες και από εκείνη την πλευρά για να αυξηθεί η δυνατότητα μεταφοράς ροών από τον νότο προς τον βορρά. Κατά τη διάρκεια πάντως της διαδικασίας του διαλόγου λοιπά, ε, δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι οι διαχειριστές, όλες οι αρχές και όλοι οι χρήστες με τη συμμετοχή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πετύχουμε αυτό που βλέπετε σε αυτήν εδώ την διαφάνεια δηλαδή η αύξηση της ροής. Έγιναν επενδύσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων και έτσι μπορέσαμε να έχουμε πέντε φορές την ε, ροή σε μεγαβάτ. Και το 2015, πολύ σύντομα δηλαδή, θα είναι πολύ περισσότερο όπως βλέπετε και στη διαφάνεια αυτή. Χρειάστηκε βέβαια να προχωρήσουν διάφορες διαδικασίες, ο ΕΣΠΕ, εξαιτία ε, των απαιτήσεων που υπάρχουν από την γαλλική νομοθεσία. Από πλευράς της Γαλλίας όμως δεν έγιναν αρκετές επενδύσεις για να διπλασιαστεί η ποσότητα μέσω νέος διαδρομής από τα Πυρηναία που να φτάνει στο 12-14 ΜΒ το χρόνο και εμπορικού λόγου και λαμβάνοντα υπόψη τοπικέ αγορέ τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία. Μάλιστα όλα αυτά όταν η οικονομική κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη ώστε οι χρήστες να είναι ε, διατεθειμένοι να κάνουν κάποιους συμβασμούς για τα πρώτα χρόνια χρήσης. Πάντως το πιο βασικό στην υπόθεση αυτή δεν έλαβε υπόψη τις εξελίξεις, δηλαδή ότι οι υποδομές αυτές βασίζονται σε ένα βασικό στοιχείο που είναι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού στα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στις διαδρομές, στις πηγές, στις περιοχές δηλαδή που προσφέρουν ενέργεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ανατολικές χώρες που ξέρω ότι σας απασχολούν επίσης. Εδώ βλέπουμε τις υποδομές που έχουν ήδη εντοπιστεί και που μπορούν να βοηθήσουν στην διασυνδετικότητα, στον τρόπο διασύνδεσης μέσω αγωγών δηλαδή και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Έχουν γίνει, όπως σας είπα, πολλές προσπάθειες έτσι ώστε οι ροές να περνάνε από τα δίκτυα των δύο χωρών είτε πρόκειται για εθνικά δίκτυα είτε για ευρωπαϊκά. Έτσι εντοπίστηκαν οι συγκεκριμένες υποδομές και το κόστος που απαιτούν για να έχουμε και μια καλή ποιότητα. Από πλευρά τη Γαλλία, σε μία από τι υποδομέ που εντοπίστηκαν και που είναι αναγκαία να φτιαχτεί για να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, είναι το ΕΝΑΝ. Που είναι σε κόκκινο και το βλέπετε πάνω δεξιά. Πρόκειται για ένα σχέδιο 200 χιλιόμετρων 1.500 εκατομμύρια εκτιμάει η γαλλική κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να ληφθεί η απόφαση πρώτα. Χρειάζεται όμως ε, διαβούλευση, κάτι το οποίο είναι λογικό, πολύ λογικό, δεδομένων των χαρακτηριστικών της υποδομής αυτής. Συνεπώς η εκτέλεση του έργου αυτού στη Γαλλία θα βοηθήσει να καλυφθεί το δίκτυο μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Κάτι το οποίο θα είναι αναγκαίο για τα επόμενα χρόνια. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές έδωσαν στη Γαλλία στα πλαίσια ενός σχεδίου ανάκαμψης 100 εκατομμύρια για να συμπληρώσει τον άξονα Βόρεια Αφρική, Ισπανία, Γαλλία. Πρέπει εδώ όμως να πούμε ότι απαιτείται και το υπόλοιπο του έργου. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα χρήματα για τον αρχικό του στόχο. Ο άξονας παντως βόρας πάντως, βόρας. η διαδρομή αυτή σύνδεσης Ισπανίας-Γαλλίας αναφέρεται και στο έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε από την έσω στην αρχή της χρονιάς που είναι ένα δίκτυο διαχειριστών ενέργειας, που αναφέρει ε, το τι πρέπει να συμπληρωθεί και αναφέρει το σχέδιο ανάπτυξης ευρωπαϊκών δικτύων μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια πλήρης ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τεχνικά χαρακτηριστικά έχοντας χρησιμοποιήσει αναλυτές και ειδικού από διάφορες πλευρές. Στο έγγραφο αυτό αναλύονται λοιπόν πάρα πολλά προγράμματα και σχέδια προκειμένου να πετύχουμε την ολοκλήρωση των αγορών. Παρατηρούμε όμως ότι αν έχουν προχωρήσει μέχρι το 2020 τα σχέδια τα οποία αναφέρονται εκεί θα υπάρχει μια τέτοια ολοκλήρωση όπου το φυσικό αέριο θα μπορεί να επεκταθεί περισσότερο. Δηλαδή το φυσικό αέριο από την Αλγερία θα μπορεί μέσω της Ιβυρικής Χερσονήσου να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γεγονός ότι υπάρχει διασύνδεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την διάθεση του φυσικού αερίου, την διαφοροποίηση της ε, ενέργειας, συνεπώς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η ενέργεια που έχει να κάνει με την διασύνδεση αυτών των ε, αξώνων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά για να λειτουργήσει αυτό, πέρα από τις υποδομές που χρειάζονται, χρειάζεται και μια αριθμιστική εναρμόνιση. Κάτι το οποίο μπορούμε να πετύχουμε μέσω των ε, κωδικών δικτύων που διαθέτει η Ένσορ και που αναφέρονται και στον κανονισμό 715. Έτσι λοιπόν, αν δείτε αυτόν το χάρτη τώρα, πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο της Κομισιόν που έχει δοθεί στη δημοσιότητα πριν από λίγες μόνο μέρες. Εδώ φαίνεται η στρατηγική ε, στάση, το top-down, αντί για το down-up. Εφόσον εντοπίσει λοιπόν, μάλλον εφόσον συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κατευθύνσεις αυτές που φαίνονται εδώ στο χάρτη και εφόσον ενισχυθεί η δυνατότητα διασύνθεσης μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, τότε δεν θα έχουμε μείνει στη θεωρία, αλλά θα έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία μπορούν να γίνουν πράξη, διότι η ισορροπία εισόδου-εξόδου είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει πολύ τις δυνατότητες ε, διάθεσης φυσικού αερίου από τη Βόρεια Αφρική. Βλέπετε τα τόξα εδώ. Είναι αναγκαία γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ισορροπία. Εγώ επικεντρώνομαι βέβαια σε αυτό το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την Ιβυρική ε, Χερσόνησο. Η διαδρομή αυτή η Ιβυρική μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση εφοδιασμού και μέσω υποδομών που ήδη υπάρχουν, υγροποιημένου φυσικού αερίου δηλαδή, και που σας έδειξα στην αρχή με το πρώτο διάγραμμα που σας έδειξα. Εμείς έχουμε έτσι κι το σχετικό εξοπλισμό. Πάντως η Βυρική Χερσόνησος είναι σαν ε, ένα στήλακα, σαν ε, μια νησίδα. Και πρέπει να βασιστούμε στο ευρωπημένο φυσικό αέριο. Και προς το παρόν, εντάξει, μπορέσαμε έτσι να αναπτύξουμε τις αγορές μας περισσότερο, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε και τις εγκαταστάσεις ε, επανεροποίησης για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Έτσι κι αλλιώς πολλοί έχουν ε, ποσοστώσεις. Η Ιβηρική Χερσόνησος πρέπει έτσι να αποτελέσει σημαντικό παίχτη στην διεθνή αγορά με διαφοροποιημένες μορφές. Αν θυμηθούμε τι γινόταν τη δεκαετία του 60 του 70 που δεν αναφέρεται εδώ στο διάγραμμα, εμείς είχαμε από την Λιβύη και ποτέ ε, ενέργεια και ποτέ δεν είχε υπάρξει διακοπή, ποτέ δεν είχε υπάρξει πρόβλημα. Εδώ και πολύ καιρό η Ισπανία ήταν η μόνη που είχε πελάτη τη Λιβύη. 40% του εφοδιασμού της ισπανικής αγοράς. Μετά υπήρχε και η Αίγυπτος. Με την κρίση όμως των τελευταίων μηνών δεν επηρεαστήκαμε για τη Λιβύη, εκεί που κόπηκε ο εφοδιασμός, ε, πρόκειτο για ε, περιθωριακές ποσότητες. Ευτυχώς υπάρχει διαφοροποίηση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι δεν πρέπει να προετοιμαστούμε στην περίπτωση που προκύψουν πιο σοβαρά προβλήματα. Και τώρα για το εγκροπημένο φυσικό αέριο. τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα και ακόμα περισσότερο στο μέλλον, όταν θα έχουμε περισσότερες ε, χώρες, θα έχει μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εδώ απευθύνομαι στον κύριο Βινουά, πρότεινε η εταιρεία μας στις αρχές, ήδη από τις αρχές του 2010 που ήταν ήρεμη η κατάσταση ακόμα, να ετοιμάσει μια τεχνική μελέτη για τις ε, συνέπειες από την διακοπή εφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η μελέτη αυτή είναι στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα της Ναγκάς. Ε, Αναφέρονται εκεί διάφορες χώρες με ποσοστά, με τα σενάρια σε περίπτωση κρίσης. Και οι συνέπειες θα είναι μικρές. Βέβαια, εννοείται ότι εφόσον υπάρχει πλήρης διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, είναι κάτι από το οποίο μπορούν να αποφεληθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που υπάρχει κάποια κρίση με διακοπή διάθεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ένα σύστημα με πλήρη διασύνθεση μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη σταθερότητα. Δεν θέλω να τελειώσω χωρίς να αναφερθώ σε κάτι άλλο, στις πηγές, στις υποδομές και στο βασικό θέμα μας που είναι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Είπαμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το φυσικό αέριο, τη σχέση του με την ε, παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά εδώ πρέπει να δούμε και τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Εδώ βλέπετε στο διάγραμμα αυτό ε, πράγματα τα οποία είναι πραγματικότητα στην Ισπανία. Βλέπετε εδώ την καμπύλη από τη χρήση των διαφόρων πηγών ενέργειας στις 9 Νοεμβρίου του 2010. Ήταν μια μέρα με ιδιαίτερο αέρα. Είναι η δεύτερη, το δεύτερο σκίτσο που βλέπετε. Καλύφθηκε περίπου η μισή, ε, οι ανάγκες κατά το ίμιση της ημέρας εκείνης. 46%. Ενώ στις 27 Αυγούστου 2009 που δεν είχαμε άνεμο, τότε χρειάστηκε βέβαια συνδυασμό με άλλες πηγές. Άρα, εφόσον υπάρχει και η ολική ενέργεια και το φυσικό αέριο και μπορούμε να περνάμε από το ένα στο άλλο ανάλογα με την ε, κατάσταση, μπορούμε να ικανοποιήσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας. Χρειάζεται ελαστικότητα λοιπόν, δηλαδή δυνατότητα τροφοδότησης ε, δυνατότητα αλλαγής από το ένα μέσο στο άλλο. Το κόστος όμως της δυνατότητας αυτής του συστήματος αναλλαγής είναι σημαντικό. Αλλά χαμηλό, αν λάβουμε υπόψη μας το συνολικό κόστος και αν λάβουμε υπόψη μας το τι πληρώνει τελικά ο χρήστης στο σπίτι του. Άμα δεν έχει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, για παράδειγμα. Η ολική ενέργεια πάντως μπορεί να βοηθήσει πολύ σε συμπλήρωμα στα δίκτυα. Όταν έχουμε άνεμο πρέπει να υποφελούμαστε από αυτόν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συμπεριλάβουμε και αυτή την πηγή ενέργειας. Αλλιώ δεν στα αρκετά από την ενέργεια που έχουμε στη διάθεσή μας στις χώρες μας. Αύξηση λοιπόν διασύνδεση, δυνατότητα διασύνδεση τη Ιβυρική Χερσονήσου με τον υπόλοιπο κόσμο. Διαφοροποίηση και ισορροπία εισόδου ενέργεια. Ολοκλήρωση των αγορών και συμπερίληψη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές πολιτικές και θεσμικές εκεί όπου αυτές λαμβάνουν χώρα. Το κόστος του διαδρόμου αυτού είναι χαμηλότερος από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις που χρειάζονται βέβαια, αλλά και σε απόλυτη τιμή, αλλά και αν λάβουμε υπόψη μας την διαφοροποίηση που μας επιτρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Τα νούμερα τα συγκρίνουμε. Είναι πολύ σημαντικά. Οι δηλαδή. Ο εφοδιασμός πρέπει να προέρχεται από διαφορετικά μέρη και μισορροπία για να μπορούμε να αποφύγουμε προβλήματα σε περίπτωση εκτακτών περιπτώσεων. Ιδιαίτερα πρέπει να φροντίσουμε την διασύνδεση με γείτονες χώρες και με χώρες με τις οποίες έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε, όπως είναι της Βόρειας Αφρικής. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι βασιζόμαστε σε σενάρια για την παρουσίαση αυτή που μόλις ε, κάναμε. Άρα υπάρχει ρήτρα αποποίησης ευθύνης και αυτό ήθελα επίσης να σας το έχω πει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Ντελαφλόρ. έχουμε ακόμα χρόνο. Μήπως ε, θα ήταν χρήσιμο να δώσουμε τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Να προχωρήσουμε αμέσως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βινουά, ο οποίος εκ μέρους της Κομισιόν ε, θα συμπληρώσει τις ε, πληροφορίες που ακούσαμε, θα μας πει ε, τι θέματα εξετάζονται εντός της Κομισιόν, ώστε κατόπιν οι συνάδελφοι να θέσουν και στους δύο μίλητες ερωτήσεις. Κύριε Βινουά, σας καλωσορίζω. Συχνά μας επισκέφτεστε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε τέτοιες ε, συζητήσεις και θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια ανεφοδιασμού του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ιδιαίτερα μετά την κρίση του Ιανουαρίου 2009. Νομίζω ότι υπάρχει κοινή συνένεση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το τι απαιτείται και είναι σαφές ότι πρέπει να ε, ζούμε με βάση την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ε, και πετρελαίου και ε, φυσικού αερίου. Η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να ισχύει, διότι με την μείωση των χωρίων αποθεμάτων μας θα πρέπει να αυξήσουμε τις εισαγωγές. Ας δούμε λοιπόν τώρα τις ε, πηγές εισαγωγών. Βλέπετε ποιοι είναι οι μεγάλοι προμηθευτές. Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος και σε, ε, και σε πετρέλαιο και σε αέριο. Αυτό φυσικά είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Και βλέπετε ότι έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση ε, στο φυσικό αέριο από ό,τι έχουμε στο πετρέλαιο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό προσεκτικά. Τα καλά νέα όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι ότι έχουμε τρεις μεγάλους ε, προμηθευτές ε, την ε, Ρωσία που παρέχει περίπου το 1 τρίτο το 23% των, της καταναλωσής μας. Η Νορβηγία είναι πολύ σημαντική. Μπορεί κανείς βέβαια να ισχυριστεί ότι η Νορβηγία είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αποτελεί μέρος λοιπόν της ευρύτερης οικογένειας μας. Συμμετέχει και στην κοινή αγορά δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η Νορβηγία είναι εξωτερικός προμηθευτής, ωστόσο είναι αρκετά αυτόνομη η Νορβηγία όσον αφορά την διαχείριση των αποθεμάτων της. Και βλέπετε την Αλγερία που είναι ο τρίτος βασικός προμηθευτής, το οποίο σημαίνει ότι η Μεσόγειος αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των, των αποθεμάτων μας. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται και γι' αυτό είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς τι θέλουμε. Θέλουμε διαφοροποίηση. Ο Τσέρτσιλ τη δεκαετία του 20 ε, έλεγε ότι ένα είναι ο κανόνα όσον αφορά το πετρέλαιο, διαφοροποίηση, διαφοροποίηση και διαφοροποίηση. Και θέλω να σα εξηγήσω ότι όταν μιλάμε για αγωγού ε, πολύ εύκολο είναι να τους ε, ιεραρχήσουμε ανάλογα με την συμβολή τους ε, στη διαφοροποίηση. Υπάρχει διαφοροποίηση της πηγής, ε, διαφοροποίηση της διαδρομής και διαφοροποίηση των, των αντίστοιχων ε, και θα σας το εξηγήσω αυτό. Έχουμε πέντε αγωγούς ε, που προμηθεύουν αέριο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον Βόρειο που είναι η Νορβηγία, έχουμε Ανατολικά τη Ρωσία, έχουμε τον Νότιο, Βόρεια Αφρική και ε, τη Βόρεια Αφρική Έχουμε το LNG που μπορεί να προέρχεται από το Τρίνιντα, το Τομπάγκο, το Κατάρ ε, και ξέρετε ότι το Κατάρ είναι ο βασικός προμηθευτής αυτή τη στιγμή και κατόπιν έχουμε τον ε, νότιο αγωγό, την νότια διαδρομή. Και το νότιο διάδρομο, <laughs> συγγνώμη. Και εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε το θέμα αυτό της διαφοροποίησης ε, και να συγκρίνουμε την κατάσταση με τον ε, αγωγό South Stream. Είναι απαραίτητο να ανοίξουμε τον ε, νότιο διάδρομο, διότι μας ε, παρέχει τα τρία στοιχεία της διαφοροποίησης. Έχουμε νέα διαδρομή, νέα πηγή. Έχουμε την Κασπία θάλασσα, όπου και ε, εδώ υπάρχει ε, τόσο φυσικό αέριο όσο υπάρχει σε όλη τη Ρωσία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πολύ να ανοίξουμε τη διαδρομή αυτή και ε, έχουμε κατόπιν το Τουρκμενιστάν, το Αζερβαϊτζάν, το το, το Ιράκ, μπορεί να έχουμε και άλλους, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι η Κάσπρο ο μόνος προμηθευτής του South Stream, έτσι, δηλαδή δεν προσθέτουμε απλά μία νέα διαδρομή, Το South Stream δηλαδή παρέχει ε, νέο αγωγό, όχι όμως νέα πηγή. Ε, πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε τα πλεονεκτήματα του νότιου διαδρόμου με το South Stream. Ε, ο στόχος μας θα πρέπει, δηλαδή, θα πρέπει να είναι να ανοίξουμε αυτόν τον νότιο διάδρομο που συχνά ονομάζεται ο τέταρτος διάδρομος. Αυτή είναι η πολιτική μας. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τι κάνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, όπως ε, πολύ σαφώς εξήγησε ο κύριος Ντελαφλόρ. Πρέπει να διασφαλίσουμε όταν ε, το αέριο εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να πάει οπουδήποτε. αυτό ε, αυτός είναι ο στόχος μας. θα πρέπει να θεωρείται το αέριο ευρωπαϊκό αέριο πια και να μπορεί να διοχετευτεί όπου είναι απαραίτητο. Τον Ιανουάριο του 2009 με την ε, κρίση του φυσικού αερίου από την ε, Ρωσία στην Ουκρανία είδαμε ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε πολύ αέριο, το οποίο όμως δεν μπορούσε να διοχετευτεί στις χώρες που επηρεάστηκαν από την διακοπή στην παροχή. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν αποθέματα ασφαλείας, ε, θα πρέπει να, έχουν, ε, να είναι αντικείμενο σωστής διαχείρισης και αυτό είναι ένα θέμα που ε, απασχόλησε και τις Ηνωμένε Πολιτείε κατά ε, την καταστροφή του ε, κυκλώνα Κατρίνα στην, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα επικεντρωθώ επασεπτώσει περισσότερο στο φυσικό αέριο, διότι αυτός ήταν ο στόχος μου και θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε την κατάλληλη υποδομή και ε, την σωστή ανταπόκριση. Ε, σωστό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση και πολιτική υποστήριξη για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Είναι κάτι που έχουμε κάνει και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια Όλα αυτά όμως ε, θα πρέπει να ε, συντονιστούν και η πρότασή μας ε, του φθινοπόρου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου θα ασχοληθεί με όλα αυτά και αυτή και αυτό είναι το, και το θέμα της έκθεσης Βάγνερ που έχει ήδη ψηφιστεί στην ε, Ήτρε και θα πάει στην Ολομέλεια νομίζω την, τον επόμενο μήνα, η οποία είναι πολύ χρήσιμη έκθεση διότι προτείνει ακριβώς αυτά που προτείνουμε και εμείς. Τα προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας υπάρχουν στη Βαλτική. Ε, έχουμε την διασύνθεση ε, ε, βορρά-νότου, έχουμε στην Ανατολική Ευρώπη και θα έχουμε και τον νότιο διάδρομο. Και χρειαζόμαστε και εξωτερική διάσταση στην εσωτερική μας αγορά. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε σωστές εταιρικές σχέσεις με τις γειτονικές μας χώρες και με τους προμηθευτές. Ο κανονισμός 994 2010 είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να εφαρμόσουμε ε, την ε, πολιτική ε, με την βοήθεια του εισηγητή του Κοινοβουλίου καταφέραμε να, περάσουμε τον, να ψηφίσουμε τον κανονισμό αυτό. Είναι κανονισμός που αντικαθιστά ε, οδηγία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως. μιλάμε για πολλές ανασφάλειες γύρω μας υπάρχει ο κίνδυνος ε, αύριο να υπάρχουν προβλήματα στην Αλγερία ή να έχουμε άλλη μια διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας. Θα είμαστε λοιπόν πιο καλά προετοιμασμένοι σήμερα από ότι ήμασταν το Ιανουάριο 2009 και μάλιστα πολύ καλύτερα, διότι Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας, και όλα τα ε, προστασίας των πελατών ε, και όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, εφαρμόσει μέτρα για να το διασφαλίσουν αυτό. Και έχουμε ζητήσει από όλα ε, τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα σε περίπτωση προβλημάτων ε, κατά την ε, παροχή, να υπάρχει συντονισμένη ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσης και αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι μπορεί να έχουμε Μπορούμε να γνωρίζουμε την ε, κατάσταση κάθε αποθέματος ε, αερίου στην Ευρώπη. Αυτό είναι αποτέλεσμα του τρίτου πακέτου. Ε, μπορεί λοιπόν να δει κανεί αμέσω τι υπάρχει από αποθέματα. Και επίσης θα αυξηθεί και η περιφερειακή συνεργασία. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι στον κανονισμό αυτόν υπάρχουν κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά την υποδομή. Έχουμε ε, το ε, ε, γνωστό πρότυπο νήμιον 1, το οποίο ανέφερε και ο κύριος Σκαρώνη Λόγω των προβλημάτων στη, Ρωσία, στη Λιβύη συγγνώμη, έχουμε τον ήμιον 1, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από άλλε πηγέ αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουν όλε οι ε, ε, σχετικέ επιχειρήσει και όλε οι χώρε ε, και θέλουμε να υπάρχει δυναμικό προ δύο κατευθύνσει σε όλε τι διασυνδέσει για να διασφαλίσουμε την σωστή παροχή σε όλου του αγωγού. Και έχουμε ένα πρότυπο προμήθεια το οποίο λέει ότι οι πελάτε θα πρέπει να προμηθεύονται αμέσω. Ε, τι γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ε, κανονισμό αυτόν. Καταρχήν κάθε χώρα θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου με όλες του ενδιαφερόμενου ε, και όσον αφορά τα αποθέματα αερίου και όσον αφορά του μεταφορεί και του μεγάλου πελάτε, ώστε να διασφαλιστεί καλή αξιολόγηση του κινδύνου και αυτό κατόπιν θα οδηγήσει σε προληπτικά μέτρα για να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι. Και επίση θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια για ε, επίγουσας σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο και για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα. Ε, όλα αυτά γίνονται αυτέ τι μέρε. Πριν τρει εβδομάδε έγινε ένα σεμινάριο σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου για να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν ε, αυτόν τον ε, κανονισμό. Ε, έχω κάποια ανησυχία ότι ίσω οι ανατολικέ χώρε δεν παίρνουν το θέμα αρκετά σοβαρά. Αλλά καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για τις χώρες αυτές, διότι πρώτον είναι οι πιο ευάλωτες, ε, είναι όμως και οι λιγότερο ευέλικτες, διότι σε μεγάλο βαθμό ε, εξαρτώνται κατά 100% ε, από έναν προμηθευτή, έχουν συστήματα τα οποία δεν είναι, με τις, δεν συμβατά με την εσωτερική αγορά και επιμένουμε λοιπόν οι χώρες αυτές ε, να κάνουν αυταπλοιακανονισμούς διότι θα είναι ζωτική σημασία για αυτές ε, ώστε να, έχουν, ε, να είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά την προμήθεια σε φυσικό αέριο. Μέχρι το τέλος της χρονιάς λοιπόν περιμένουμε την αξιολόγηση κινδύνου και τα προληπτικά σχέδια δράσης. Είναι επίσης σημαντικό στο πνεύμα αλληλεγγύης να υπάρχει ανταλλαγή των αξιολογήσεων κινδύνων μεταξύ γειτονικών χωρών διότι ο κίνδυνος, ε, ε, η αξιολόγηση κινδύνου δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένα κράτος μέλος μόνο του, πρέπει να λάβει υπόψη και το τι γίνεται στις γειτονικέ χώρες. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω πόσο μας ε, έχει βοηθήσει το πρόγραμμα ενέργειας, το Energy Program for Recovery. Θα θυμάστε ότι 4 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να στηριχθούν οι υποδομές αυτές. Όπως βλέπετε πάνω από το μισό του ποσού αυτού ε, έχει ε, δοθεί για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το ε, αέριο, κυρίως όμως στο αέριο. Και βλέπετε εδώ κάποια προγράμματά μας. Κύριε Μεσάρος, ε, παραπορεθήκατε για ε, την ε, κατά 100% εξάρτησή σας από τη Ρωσία. Μπορείτε όμως αύριο να έχετε φυσικό αέριο από την Αυστρία, διότι στο Baumkarten έχουμε ένα, ένα σύστημα reverse flow, αντίστροφης ροής. Έτσι λοιπόν... Είναι δυνατόν να αντιστρέψει κανείς τη ροή στον αγωγό από τη Ρωσία μέχρι την Ιταλία στο Baumgarten ώστε να, να μπορεί να μεταφερθεί στην Σλοβακία αέριο. Αυτό έχουμε χρηματοδοτήσει με το πρόγραμμα αυτό και είδαμε και τα προγράμματα της Ισπανίας. Χρηματοδοτούμε την Γαλλική-Ισπανική Διασύνδεση και ενισχύουμε και την γαλλική αγορά όσον αφορά τη διασύνθεση προς τον Νότο αλλά και προς τον Βορρά. Όλα αυτά λοιπόν πραγματοποιούνται. Βλέπετε ότι έχουμε επενδύσει πολλά στις ανατολικές χώρες ε, για να διασφαλίσουμε ευελιξία του συστήματος ε, και να ε, διασφαλίσουμε τη διασύνδεση ε, αυτή τη στιγμή. Ε, αντιμετωπίζουμε ακόμα κάποια προβλήματα στη Σλοβακία, αλλά το εξετάζουμε το θέμα. Στόχος είναι λοιπόν να υπάρχουν διασυνδέσεις με τις χώρες αυτές. Έτσι λοιπόν βελτιώνουμε την ασφάλεια αναφοδιασμού για τις χώρες αυτές. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες και αυτό θα είναι το αντικείμενο πρότασής μας ε, στο τέλος της χρονιάς. Υπάρχει μια σειρά προτεραιοτήτων που αφορούν διαδρόμους. Ε, πρέπει να κοιτάξουμε τις διάφορες περιφέρειες, να δούμε πού είναι τα ε, αδύναμα σημεία, να δούμε όμως και πού είναι τα ισχυρά σημεία. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τα ισχυρά σημεία για να μειώσουμε ε, τα αδύναμα σημεία, να ελαττώσουμε τα αδύναμα σημεία. Για παράδειγμα, στην Βαλτική βλέπετε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τις σωστές διασυνδέσεις για το ηλεκτρικό και για το αέριο, ώστε οι τρεις βαλτικές χώρες αλλά και η Φιλανδία να ε, έχουν σωστές διασυνδέσεις με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, έχουμε την, ε, την διασύνδεση βορρά-νότου για το αέριο αλλά και για το φυσικό αέριο. Είναι κάτι που συνδέει τις χώρες των Βαλκανίων και με την Πολωνία ε, ώστε όλες ε, οι χώρες αυτές να μπορούν να, πάρουν, να λάβουν αέριο LNG, ε, υγροποιημένο δηλαδή φυσικό αέριο, η οποία είναι η πιο, η πιο σίγουρη πηγή ενέργειας. Επίσης, συνεχίζει να είναι σημαντική προτεραιότητα ο νότιος διάδρομος. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να ανοίξει αυτός ο νότιος διάδρομος. Όπως βλέπετε, είναι κάτι που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Ανατολική Μεσόγειο, τις πιθανές πηγές αερίου για το μέλλον. Μιλώ για την Κύπρο, το Ισραήλ και το Λίβανο. Ξεκινάμε συζητήσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, συνδέσουμε τις ε, πηγές ε, αυτές αερίου που δεν είναι καθόλου μικρές. Το Ισραήλ δηλαδή έχει 7 φορές την ετήσια κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε επιπλέον διαφοροποίηση όσον αφορά τις πηγές ανεφοδιοσμού. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο εξετάζουμε. Έχουμε ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ενδιαφέρει την Κύπρο και την Ελλάδα που ε, θα είναι ε, οι χώρες εισόδου του αέριου αυτού. Ε, έχουμε λοιπόν πολλέ πιθανέ πηγέ. Δεν σας μιλώ καθόλου για το αέριο από διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα βρίσκεται υπό ανάπτυξη, αφορά το μέλλον μετά το 2020. Θα το έχουμε βέβαια κατά νου. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες προτάσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς για να δείξουμε πώς, μπορούμε, πώς πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις υποδομές πώς πρέπει να συνεργαστούμε με τους νομοθέτες ε, και με τους άλλους ενδιαφερομένους ε, για να ε, δούμε πώς θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις και θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να έχουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν οι επενδύσεις αυτές και υπόθηκε σαφώ σήμερα πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση, το οποίο σημαίνει ότι μερικέ φορέ χρειάζεται να έχει κανεί εντό αγωγικών περιττή υποδομή, κάτι που δεν αρέσει στην ε, αγορά. Θα πρέπει να επενδύσουμε στι υποδομέ, δηλαδή μερικέ φορέ είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερε υποδομέ από ό,τι φαίνεται ότι χρειαζόμαστε. Ε, έτσι λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά και να βελτιώσουμε την ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι απαραίτητα απαραίτητα γι' αυτό. Θα κλείσω λοιπόν εδώ, διότι νομίζω ότι είπα αρκετά. Νομίζω ότι και οι τρει ε, ομιλίε ε, σήμερα το πρωί όλε ε, ακολουθούσαν την ίδια κατεύθυνση και σα έδωσαν μια εικόνα σχετικά με το τι γίνεται και το τι πρέπει να γίνει. Νομίζω όμω ότι η κατεύθυνση για την ασφάλεια του ελευθεριασμού είναι σαφή. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βινουά. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η προσθήκη αυτής της ε, παρουσιάσης ε, που ακούσαμε από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή ε, ακούσαμε την πλευρά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Εσείς αναφερθήκατε σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. μη Βρήκα πολύ χρήσιμες ε, τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, ε βλέπω ότι διάφοροι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους όσοι πήραν το λόγο. Πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνομαι πολύ περίεργα. Μια που μιλάμε για χώρες, για λαούς, οι οποίοι τόσο δύσκολα έδιωξαν δικτατορίες, προσπαθούν να οργανώσουν την δημοκρατία τους και νιώθω ότι μιλώντας για τη δικιά μας ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας, ε, δείχνουμε να είμαστε εγωιστές. Πρώτον, πρώτη παρατήρηση για την διασύνδεση και για την ανάγκη να επενδύσουμε. Όντω, χρειάζονται επενδύσει, πρέπει να έχουμε τέτοια σχέδια. Συμφωνώ. Πώ όμω βλέπετε εσεί την ε, σχέση ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και πώ βλέπετε εσεί να οργανώνουμε την ιδιοκτησία ε, υποδομών. Πώ ξέρουμε τι ανήκει σε ποιον. Πώ το οργανώνουμε αυτό με τις επιδοτήσεις, γιατί το Ναμπούκο είναι ιδιωτικό. Πώς θα οργανώνουμε όλα αυτά. Δεύτερον, μήπως θα έπρεπε να περάσουμε σε μία σχέση εταιρική επενδύσεων για τα φωτοβολταϊκά και λοιπά με την νότια πλευρά της Μεσογείου. Και τρίτον, όσον αφορά το γεωπολιτικό στοιχείο, γνωρίζω καλύτερα τα θέματα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τις χώρες αυτές νοτίως της Μεσογείου μας λένε ότι η Αφρική αναπτύσσεται αυτόνομα και ότι κάποια στιγμή θα χρειάζεται ενέργεια και άρα θα έχει γεωπολιτικές συμφωνίες με τις χώρες ε, αυτές της Βόρειας Αφρικής. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος ε, Ματορέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βινουά σε σχέση με κάτι που είπε και ο κύριος Δελαφλόρ. Γιατί βλέπετε ότι θεωρούμε προτεραιότητα να ενισχύσουμε τον άξονα Αφρική, Ισπανία, Γαλλία. Χρειάζονται χρήματα για να αναπτυχθεί η διασύνδεση αυτή και μέσω της Καταλωνίας. Και μια που μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη αυτή, ξέρουμε ότι υπάρχει και το σχέδιο Μεριντάν. Είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά από ό,τι είπε ο κύριος Ντελαφλόρ, η Γαλλία, το Εριράν, το έχει ξαναξεκινήσει. Ρωτάω λοιπόν, μπορεί αυτό να ενισχύσει τον άξονα Αλγερία-Ισπανία-Γαλλία, μια από αυτός είναι ο στόχος, αν δεν έχουμε και τον αγώ φυσικό αερίο ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Φαντάζομαι ότι μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να επανεργοποιηθεί θα πρέπει να επανεργοποιηθούν και άλλα πράγματα. Τώρα μια που σας έχουμε εδώ, θέλω να ξέρω γιατί δεν λειτουργήσαν μέχρι τώρα αυτά. Παλιότερα είχαμε μιλήσει για το κόστος, για διαφωνίες μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Αλλά υπήρχε και κανένα άλλο πρόβλημα. Και τέλος θέλω να ζητήσω ένα στοιχείο από τον κύριο Τελαφλόρ. Αναφέρθηκε στο τι μπορεί να κάνει η Ιβυρική Χερσόνησος για να αποφύγουμε προβλήματα σε περίπτωση διακοπής προβλημάτων όπως είχαμε τη Ρωσία και την Ουκρανία. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη μας τις διάφορες παροχές, φυσικό αέριο, υγροπημένο κτλ. Τι όγκο μπορεί να προσφέρει ο διάδρομος αυτός προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πόρτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, άκουσα σήμερα το πρωί και θυμήθηκα το γερμανικό θεατρικό έργο «Gas», φυσικό αέριο, που μιλά για την κοινωνία και την τρέλα της με την παραγωγή φυσικού αερίου. Μήπως όμως πρέπει να έρθουμε στην πραγματικότητα. Αν θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που το χρησιμοποιούμε σήμερα το φυσικό αέριο, δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του πλανήτη κατά δύο βαθμούς μέσα σε αυτόν τον αιώνα και ούτε και θα αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού εκτός Ένωσης και πιθανότατα δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα πολιτικής ε, καταπίεσης στις χώρες που μας προμηθεύουν το φυσικό αέριο. Μόλις πέρσι είδαμε τη δημοσίευση του δικού χάρτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα μέχρι το 2050 που εμπνεύστηκε από τον οδικό και ενέπνευσε μάλλον τον οδικό χάρτη της Κομισιόν για φέτος που είδαμε σαφή επέκταση στις ε, ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Δηλαφλός μας είπε σε μια ε, μέρα με πολύ αέρα μπορεί να παράγει το μισό της ενέργειας που χρειάζεται η Ισπανία. Θα μπορούσε το υπόλοιπο μισό να το παράγει μέσω της θερμικής ενέργειες. Είδαμε ήδη από, τη Μαρό, από το Μαρόκο και από τη Σενεγάλη ότι η συμπυκνωμένη ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με την αιωλική ενέργεια από την Ιρλανδία μέχρι και την Εστονία, πράγμα που ήδη συζητείται από τους υπουργούς μας, θα μπορέσουμε όντως να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία για να συγχρηματοδοτήσουμε κινείται μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το φυσικό αέριο μόνο να συμπληρώνει τα κενά. Νομίζω λοιπόν ότι αν τα κάνουμε όλα αυτά θα πρέπει να βασιστούμε στον ηλεκτρισμό και στα smart grids και όχι στο φυσικό αέριο και τα δικά του smart grids. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη των, ε, του εισηγητή γι' αυτό. Ο συνάδελφος Τούρμας, σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις στον κύριο Τελαφλόρο. Μια ναι, για τους διαδρόμους Ισπανίας-Αλίας. Είπατε πως υπάρχουν κάποια προγράμματα που ετοιμάζονται. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα. θα, ποια θα είναι η χωρητικότητά τους όταν ολοκληρωθούν. Και βλέπετε εμπόδια στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Δεύτερον, σας ευχαριστώ για την πιο ισορροπημένη εικόνα που μας δώσατε για τη σχέση μεταξύ φυσικού αερίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, ε, στον κύριο Σκαρόνη είδαμε πολύ ιδεολογικά, ε, μάλλον εξειδανικεύει την κατάσταση. Όταν μιλάμε για αποθήκευση φυσικού αερίου, χρειαζόμαστε περισσότερη ταχεία αποθήκευση. Και ποια είναι η απόψή σας για τις αγορές ηλεκτρισμού intraday. Μια παρατήρηση επίσης για τον κύριο Βενουά και με βάση το όσα είπε ο κύριος Βότσον. Πιστεύω πως η Κομισιόν θα πρέπει να εξισορροπήσει το θέμα. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση που θα υπάρξει μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα είναι η επάρκεια στην ενέργεια και οι ανανεώσιμες. Τόσο κάνουμε στο φυσικό αέριο είναι σημαντικά, αλλά στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων σίγουρα ακολουθεί τις προσπάθειες πρέπει να κάνουμε για την, για την ε, επάρκεια και το φυσικό αέριο. Είπατε ότι ο Ναμπούκο θα πεθάνει γιατί δεν έχει παραγωγούς μέσα στους ε, μετόχους του. Από την άλλη πλευρά η Κομισιόν είναι πολύ αισιόδοξη για τον Ναμπούκο. Ποιο είναι το επιχείρημα του κ. Σκαρόνη ότι μόνο καταναλωτέ υπάρχουν από την πλευρά του αγωγού Ναμπούκο. Είναι σε αυτό σοβαρό πρόβλημα για την άποψή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους δύο συγητές πρώτα απ' όλα και τον κύριο Σκαρόνη βέβαια που μίλησε πριν. Πολύ σύντομα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τελαφλόρ. Μπορεί να μας εξηγήσει με τι όπλα σκοπεύει η αναγκάς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ε, αντίθεσης των πληθυσμών αλλά και των ε, αρχών της Ισπανίας και των αυτόνομων ε, περιφερειών και των δήμων και ποια είναι η θέση της αναγκάς στο πρόβλημα αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Σκαρόνη όσον αφορά τις μη συμβατικές ε, πηγές, σχιστόλιθο για παράδειγμα. Και μια ερώτηση τώρα προς τον κύριο Βινουά για την επιλογή ε, προγραμμάτων υπέρ της Ευρώπης. Η Κομισιόν τι θέση θα υιοθετήσει για να προωθήσει τέτοια προγράμματα ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή συνοχή δηλαδή να έχουν κάποιο ευρωπαϊκό στοιχείο, να συμφέρουν την Ευρώπη. Διότι εγώ βλέπετε υπέβαλα μια έκθεση στην Επιτροπή αυτή και θα ήθελα να μου πείτε γιατί έχει σχέση με αυτή. Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στον κύριο Ντελαφλόρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας με τη σειρά. Για τον κύριο Ντί. Αναφερθήκατε στο δημόσιο τομέα και τις επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις υποδομές, τις επιδοτήσεις και πώς οργανώνονται όλα αυτά. Όπως είπα και στην αρχή, από τη στιγμή όπου υπάρχει μια δέσμευση με τον ρυθμιστή, ώστε υποδομές να κατανέμονται με λογικό τρόπο, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τις επενδύσεις που χρειάζεται. Το κόστος της χρηματοδότησης είναι ένα χαμηλό κόστος, πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα και οι υποδομές να κοστίζουν λιγότερο και άρα οι επιπτώσεις στη συνέχεια είναι χαμηλές. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν εξαίρετα από τον ιδιωτικό τομέα, άπαξ και υπάρχει φυσικά δέσμευση από πλευράς των ρυθμιστικών αρχών, γιατί πιστεύουμε ότι μία υποδομή φυσικού αερίου είναι για 40-50 χρόνια. Και ξέρουμε τη σχέση που υπάρχει, και απαντάω τώρα και στον κύριο Τουρμές έτσι, ότι το φυσικό αέριο δηλαδή μπορεί να είναι μια μεταβατική ενέργεια, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο απόσβεσης έτσι ώστε το κόστος να είναι χαμηλό. Οι ιδιωτικέ εταιρείε όπως η δικιά μας είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τέτοιου είδου επενδύσεις. Και περνάω την ερώτηση της κυρίας Μαντουρέλ. Ναι, είμαστε όντως επιχείρηση που ασχολείται ιδιαίτερα με τις υποδομές. Δεκαετίες ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα. Υπάρχει ρυθμιστής πίσω από μας και τα προγράμματά μας είναι προγράμματα υψηλής ποιότητας, με προδιαγραφές ποιότητας δηλαδή αντίστοιχες τουλάχιστον με εκείνες βάσει των οποίων λειτουργούν άλλε άλλες χώρες. Υπάρχει δε και απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία μας και το ξέρουν και άλλοι διαχειριστές οι οποίοι λειτουργούν με ένα κόστος που πολύ συχνά είναι 30, 40, 50, ακόμα και 100% μεγαλύτερο από το δικό μας. Αναφερθήκατε στην αντίσταση του τοπικού πληθυσμού. Ναι, αλλά... Η οικοδομή, η οικοδόμηση μάλλον ενό αγωγού γίνεται με κάποιες προμήθειες και σας είπα ότι το κόστος είναι χαμηλό. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ειδικευμένες όπως είναι η δικιά μας φροντίζουν οι υποδομές τους να κατασκευάζονται με ανταγωνιστικές τιμές. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνει την ύφη γι' αυτό τελικά ο τελικός χρήστης. Όχι. Γιατί δεν προχωρήσαμε περισσότερο. Είπα ότι ευτυχώς τα 4-5 χρόνια που έχουμε δουλέψει έχουμε πετύχει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε από το 0 και λέμε ότι το 2015, πολύ σύντομα δηλαδή, θα έχουμε αυξήσει κατά πολύ την ε, χωρητικότητά μας, τις δυνατότητες μεταφοράς. Πρέπει να δούμε τι γίνεται γενικότερα στην αγορά. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει μια ημερίδα διαλόγου Γαλλίας ε, Ισπανίας και ο πρόεδρος Λακρέ είχε πει κοιτάξτε για θέματα υποδομών δεν είναι μόνο η αγορά που βάζει τους κανόνες. Φανταστείτε αν έπρεπε έτσι να γίνει ο πύργος του Άιφελ ή το ιδιόρυγα του Σουέζ. Γι' αυτό λοιπόν και από στρατηγικής πλευράς φυσικά και πρέπει να δούμε πρώτον τι βγαίνει και δεύτερον σε μια περίοδο όπως είναι η σημερινή πως η Ισπανία και η Γαλλία μπορούν να ζητήσουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις από πλευράς της αγοράς. Και τέλος να δούμε κατά πόσο το κόστος και οι τελικές επιπτώσεις του είναι τόσο μεγάλες ώστε το οικονομικό βάρος να είναι τέτοιο που να μην μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να το αναλάβουμε. Είμαι πάντως πεπισμένος και ελπίζω ότι μετά από αυτή τη συζήτηση να συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμεύεται μακροπρόθεσμα και να μην χρειάζεται να περιμένουμε το 10, το 5, το 2. Τώρα, το μισό του διαδρόμου έχει ήδη ξεκινήσει. Γιατί Απλώς διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να γίνει, ήταν ανάγκη, χρειαζότανε. Το σύνολο του διαδρόμου Αφρικής, Ισπανίας, Γαλλίας ε, θα ήταν λογικό να αναπτυχθεί παρετέρω. Οι δυνατότητες φυσικού αερίου που μπορεί να μπει και να κυκλοφορήσει και να συνεισφέρει όπως και η Δυτική Χερσόνησος στο μέλλον ε, της ανεξαρτησίας εφοδιασμού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ σήμερα. Μπορούν έτσι να προσθεθούν περισσότερα μεγαβάτ. Και με το υγροποιημένο φυσικό αέριο επίσης μπορούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες. Γιατί κάθε φορά μιλάμε για 10 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν είναι πολύ. Τέλος για τον κύριο Σώσα. Ο ιβυρικός διάδρομος. Σας είπα ποια είναι τα εμπόδια. Αλλά το βασικό ίσως είναι η συνεννόηση μεταξύ των ατόμων πώς ε, θα συμβιβάσουμε διαφορετικές νοτροπίες. Και σιγά σιγά ξεπερνιέται αυτό το εμπόδιο τα τελευταία χρόνια. Το απαιτεί αυτό ο στόχος του 2015, τη συνεργασία μεταξύ μας. Για τις υποδομές, για να υπάρχει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό αέριο ή τέλο πάντων προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα το φυσικό αέριο ανάμεσα στη σημερινή κατάσταση και την μελλοντική, όπου θα χρησιμοποιούμε εναλλακτικέ ενέργειες, χρειάζονται υποδομές. Και ας είναι υποδομές το μικρότερο μέρος του κόστους, χρειάζονται μεγάλες υποδομές με ελαστικότητα. Και ακριβώς σε αυτές οι καταστάσεις επανεροποίηση είναι και ο πιο ευέλικτος εξοπλισμός και υποδομή που χρειαζόμαστε. Επενδύσεις στις υποδομές για το φυσικό αέριο χρειάζονται έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν θέλουμε να αναπτύξουμε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θέλω να πω στον κύριο Σώσα, ναι, ότι η Ισπανία ευτυχώς Είμαστε έτη φωτός μπροστά όσον αφορά το ίμπι, τζίμπι και μπίμπι. Η Ισπανία έχει προχωρήσει πολύ όσον αφορά τις εγκαταστάσεις επανεροποίησης. Πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις ορισμένες ε, περιοχές όπου αντιμετωπίζουμε προβλήματα άδεια, έχουμε καθυστερήσεις. Γι' αυτό και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά αν συγκρίνουμε τι γίνεται σε εμά και αλλού, το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Τέλος, το μη συμβατικό αέριο. Εμεί δεν έχουμε τίποτα. Έτσι κι εξαρτώμεθα πλήρως, συμβατικό ή μη συμβατικό. Αλλά βέβαια και η εμφάνιση και η ανάπτυξη μη συμβατικού αερίου στις ΗΠΑ είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις στο κατά και αλλού και ότι πολλές χώρες ε, το σκέφτονται και προβληματίζονται. Σχιστόλιθου κλπ. Το υγροποιημένο, το οποίο αρχικά ήταν στι Πολιτείε έφτασε στις χώρες μας. Οπότε το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Με τέτοιες πηγές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο απαιτεί εγκαταστάσεις που εμείς μπορούμε να θέσουμε στη διάθεση της υπόλοιπη Ευρώπης. Είναι δύσκολες αυτές οι εγκαταστάσεις. Εμείς τις έχουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις εγκαταστάσεις που ήδη διαθέτουμε και να φροντίσουμε για την διασύνδεση. Αυτή να αναπτύξουμε παρετέρω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βινουά. Εγώ συμφωνώ με το όσο είπε ο κύριος Οντί, ότι δηλαδή είναι κάπως ε, εγωιστικά όλα αυτά και ότι δεν καλύπτουν ε, όλα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κομισιόν ε, σε εταιρικέ σχέσεις για να αντιμετωπίσουμε την ενέργεια. Σίγουρα δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, θέμα αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Η συνεργασία με την Βόρεια Αφρική, με τις χώρες του Περσικού Κόλπου θα πρέπει να πω ότι δεν έχουν εκφράσει μεγάλη ε, ενδιαφέρον για να συνεργαστούν μαζί μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Πίμπαλξ που είναι τώρα δε επίτροπος για την ανάπτυξη αφού έχει διατελέσει επίτροπος για την ενέργεια έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα που πραγματικά εξετάζει την πρόσβαση στην ηλεκτρισμό για τους Αφρικανούς, να αναπτύξει δηλαδή τους καλύτερους δυνατούς, τις καλύτερες δυνατές υποδομές στην Αφρική για να το εξασφαλίσει αυτό γιατί είναι πραγματικά πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν πως Ε, θα έχετε την ευκαιρία να το συζητήσετε, γιατί από ό,τι κατάλαβα γύρω στο Σεπτέμβριο θα ε, το προτείνει αυτό. Τώρα, για την ε, αγορά φυσικού αερίου, Πιστεύω πως ε, το θέμα είναι, ε, είναι υπό εξέταση, γίνονται προτάσεις για τη μεταφορά του φυσικού αερίου για τον ηλεκτρισμό, είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχετε κάθε είδους ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πάντως πρόκειται για μια, ένα τομέα όπου λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον ε, των πολιτών τα αποθέματα επίσης ε, ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για την κυρία Μαντουρέλ να πω για το προσχέδιο Εριντάν. Χάρη στα χρήματα του προγράμματος ανάκτησης μπορέσαμε να πείσουμε τους Γάλλους να προχωρήσουν με το Εριντάν παρά από την αρνητική ε, κατάσταση. Γιατί μπορέσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλουμε τα χρήματα στο τραπέζι και να πούμε ορίστε, προχωρήστε το Έρινταν είναι η βάση για την διασύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας για να γίνει και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί αυτό είναι μεγάλη προτεραιότητα για μας. Για τον κύριο Βότσον να πω, αν δεν είναι πια εδώ, Νομίζω πως υπάρχει μια σημαντική πτυχή στο, για το φυσικό αέριο που είναι η απελευθέρωση του από το διοξίδιο του άνθρακα. Πιστεύω πως υπάρχει, γίνεται μεγάλη έρευνα για το θέμα αυτό. Ο κύριος Τούρμες είπε ότι ναι, το φυσικό αέριο θα είναι ακόμα για 10-15 χρόνια και θα συνεχίσει να υπάρχει εφόσον καταφέρουμε να αφαιρέσουμε το διοξίδιο του άνθρακα και από ό,τι ξέρω αυτό θα δείτε όμως ότι η ανανεώσιμη ενέργεια και το φυσικό αέριο συμβαδίζουν. Μακάρι να γινόταν ο ηλεκτρισμός από τον αέρα μόνο, μια ωραία μέρα, αλλά όταν δεν υπάρχει αέρας θα πρέπει να μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι άλλο η παραγωγή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο είναι δύσκολη. Αυτές τις εγκαταστάσεις τι θα κάνουν, θα λειτουργούν κάποιες ώρες την ημέρα. Υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα εδώ που πρέπει να λυθεί για να εξασφαλιστεί σωστός συντονισμός ανάμεσα σε όλα αυτά. Τώρα για τον κύριο Τούρμες. Και τη στρατηγική 2020, της οποίας αναπόσπαστο τμήμα είναι η επάρκεια. Θα έχουμε πολύ δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις νομίζω Για το θέμα του Ναμπούκο, ο κ. Καρόνι είπε ότι το Ναμπούκο δεν έχει... Ότι μάλλον αυτό εξαρτάται από τους καταναλωτές του φυσικού αερίου και το πρόβλημα του Ναμπούκο είναι να υπάρχει μια σύμβαση για την παροχή του αερίου. Και το καλύτερος τρόπος για να το εξασφαλίσουμε αυτό είναι να έχουμε μια σύμβαση με τον παραγωγό Αζερβαϊτζάν, Τουρκουμενιστάν, Ιράκ. Όλα αυτά σίγουρα θα βελτίωναν τις βελτιώσεις. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα έγιναν πολύ σημαντικές ε, συζητήσεις για τον νότιο διάδρομο με το Αζερβαϊτζάν και με το κονσόρσιο του Ναμπούκο. Κινούνται τα πράγματα δηλαδή, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πρώτος προμηθευτής είναι ο, το Αζερβαϊτζάν. είναι ο πρώτος προμηθευτής του Ναμπούκο. Το Ναμπούκο όμως είναι κάτι το νέο, είναι ένας νέος αγωγός που διασχίζει την Τουρκία, ενώ το TGI συνδέει με την Ιταλία. Είναι συμπληρωματικά λοιπόν αυτά τα προγράμματα και νομίζω πως ο χρόνος θα δείξει ότι είναι θετική η συνεργασία μεταξύ τους. Είδαμε τι προτείνεται εδώ στις εκθέσεις. Νομίζω όλα αυτά τα κριτήρια είναι... κινούνται προς την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει ανάλυση κόστος ωφέλειας και θα πρέπει εδώ να μπουν και οι συνιστώσεις της ασφάλειας ανεφοδιασμού ή της πιθανής μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου. Είναι σαφές ότι σε χώρες ε, όπου ο Γκάσπρομ είναι ο μοναδικός προμηθευτής, αν δημιουργηθεί διασύνδεση που θα φέρνει αέριο και απαλού, φυσικά αυτό θα βοηθήσει, θα βελτιώσει την διαπραγματευτική θέση της ε, χώρας ε, στις διαπραγματεύσεις για την τιμή με την Gazprom. Και γι' αυτό και πρέπει να δούμε όλα αυτά τα ωφέλη Αυτό το κάνουμε αυτή τη στιγμή, το εξετάζουμε και θα το δείτε και στις προτάσεις που θα κάνουμε αργότερα στο το φθινόπωρο. Κυρίες και κύριοι, τις προτάσεις από μένα για να κλείσω και κατόπιν θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Αλπερτίνη. Πρώτον, ήταν πολύ χρήσιμο που είχαμε αυτήν την κοινή ακρόαση, κοινή για τις δύο επιτροπές μας. Ε, δεύτερον, να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας, βοηθήσατε πάρα πολύ. Και τρίτον, όποιος ήταν παρόν ε, και άκουσε αυτά που υπόθηκαν, κατάλαβε την πολυπλοκότητα των θεμάτων αυτών. Δεν υπάρχει απλή απάντηση στα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να έχουμε διαφοροποιημένες ε, απαντήσεις ε, στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλπερτίνη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μόνο εσά, συνάδελφε Ρόιλ, για την εξαιρετική μας συνεργασία και για το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι και οι συνάδελφοί μας έτσι γνωρίσαμε εις βάθος τα θέματα με την εμπειρογνωμοσύνη των ομιλητών μας. Να πω μόνο ε, μερικά δευτερόλεπτα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βινουά μετά την πρόταση του κύριου Σκαρόνη. Ποιες πιθανότητες μπορούν να υπάρχουν για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής αφιερωμένης στην ευρωπαϊκή διασύνδεση για να δούμε την καλύτερη οργάνωση και κατανομή διανομή μάλλον του φυσικού αερίου, που είναι ένα από τα σημεία κλειδιά που υπογραμμίσατε κι εσείς. Έχουμε την οργάνωση που μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα, που είναι η ΕΝΣΟΚ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τους ε, φορείς ε, διανομής φυσικού αερίου, αυτό έχει δημιουργηθεί μέσω της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς. Έχουμε προβλέψει, την έναρξη ισχύω αυτών των οδηγιών. Συνεργαζόμαστε δηλαδή και είμαι πεπισμένος ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε μια πραγματικά καλή οργανωμένη, ένα καλά οργανωμένο δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πλήρη χρήση και αξιοποίηση των υποδομών ηλεκτρισμού και, και φυσικού αερίου. Και γι' αυτό και πρέπει να πιέσουμε για όλη αυτή τη διαδικασία γιατί είναι κάπως επίγον να δημιουργηθούν αυτές οι οι υποδομές. Δεν μπορούμε δηλαδή να το καθυστερήσουμε. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με τους ευρωπαϊκούς στόχους και είμαι πεπισμένος ότι όλοι αυτοί αν συνεργαστούμε, θα πετύχουμε τους στόχους. Είμαι λοιπόν ε, σίγουρος πως το μέλλον είναι λαμπρό μπροστά μας.